Mes chers collègues, bonjour ou rebonjour. Allez, on... Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε εκ νέου τις εργασίες μας. On y va Allez, notre commission a décidé d'organiser... Αποφασίσαμε να οργανώσουμε λοιπόν σήμερα και αύριο μία δημόσια ακρόαση για το πακέτο σχετικά με την κινητικότητα. Αυτή η δημόσια ακρόαση θα χωριστεί σε δύο μέρη. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στις τέσσερις νομοθετικές προτάσεις που έχουν να κάνουν με την εσωτερική αγορά και τις κοινωνικές πτυχές, ενώ αύριο θα εξετάσουμε τις προτάσεις που σχετίζονται με τα διόδια. Η αγορά των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων είναι κρίσιμη σημασία για την ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία, χρειαζόμαστε έναν τομέα μεταφορών βιώσιμο, ισχυρό, σταθερό, που να παρέχει επαρκείς, επαρκείς δυνατότητες ε, ε μεταφοράς ε, και παράδοσης ε, εμπορευμάτων εντός της αγορά. αγοράς. Ο στόχος μας, όλων εδώ, είναι να εξασφαλίσουμε ότι η νέα νομοθεσία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βελτιώσει την ζωή των εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών και πρέπει επίσης να βοηθήσουμε όλους όσους ε, θέλουν να δραστηριοποιηθούν ε, στον τομέα αυτών, σεβόμενοι πάντα τους υπάρχοντες κανόνες βέβαια. Έτσι λοιπόν τα ζητήματα που φέρουν την αγορά αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα θα πρέπει να εξεταστούν από κοινού για να φτάσουν σε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα λαμβάνοντα υπόψη την προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμφερόντων των πολιτών. Το Κοινοβούλιο έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο εδώ να παίξει για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και διαπιστώνω ότι αυτή η συνεισφορά σήμερα και αύριο θα μας βοηθήσει ε, να διαμορφώσουμε αυτή τη νέα νομοθεσία προς το καλύτερο. Λοιπόν, να σας παρουσιάσω τώρα τους ε, ομιλητές σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας καλωσορίζω εδώ. Καλώς ήρθατε. Εσείς είστε εμπειρογνώμονες ε, σήμερα το απόγευμα σε αυτό το πάνελ. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Σίπερ, λοιπόν, ο οποίος είναι γενικός εκπρόσωπος της Eurocontrol Route, Καλώς ήρθατε. Η κυρία Μπερτελό, η οποία είναι εκπρόσωπος της ε, Εθνικής Ομοσπονδίας Οδικών Μεταφορών, ο κύριος Παρίγιο, πρόεδρος ε, του Τμήματος των Οδικών Μεταφορών της ε, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών. Δεν είστε μόνος εδώ βέβαια, υπάρχει μια ολόκληρη αντιπροσωπεία μαζί σας, με σημαίες, αλλά δεν θα βγάλουμε σημαίε τώρα εδώ, έτσι. Καλώς ήρθατε πάντως. Ο κύριος Λάισκο, διευθυντής ε, μιας ουγγρικής εταιρείας μεταφορών και υποστήριξης. Ο κύριος Πολόνιο αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Οδικών Μεταφορών της Πορτογαλίας, ο κύριος Βίλιατσεν, ε, πρόεδρος του Δανέζικου Συνδικάτου 3F Transport και τέλος ο καθηγητής Μπορκόφσκι από το Πανεπιστήμιο του Γκτάνσκ. Καλά το είπα. Του Γκτάνσκ στην Πολωνία. Καλώς ήρθατε. Βεβαίως ε, θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα εδώ. Λοιπόν, σας το λέω από τώρα, ευθύς εξ αρχής. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή στο ζήτημα του χρόνου. Ανυποχώρητη. Επτά λεπτά θα έχει ο καθένας. Επτά λεπτά παρέμβασης. Και Στη συνέχεια θα έχουμε τις ερωτήσεις. Μετά και τις 7 παρουσιάσεις. Για τη συζήτηση θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του ping-pong, όπως την λέμε. Δύο γύροι ερωτήσεων προς τους εμπειρογνώμονες. Στον πρώτο γύρο θα, μιλήσουν, θα μιλήσει πρώτα ο εισηγητής και στο δεύτερο γύρο τα μέλη που θέλουν το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω εδώ τους, ε, τον χρόνο ομιλία σας και αυτόν θα πρέπει να σεβαστείτε, Αγιώ θα σας κόβω το μικρόφωνο. Θα σας παίρνω το μικρόφωνο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Ισμαήλ Ακτούν, Μόνο μία παρατηρήση, αν μου επιτρέπετε, μία πρόταση δηλαδή για να διαμορφώσουμε πιο αποτελεσματικά τη συζήτησή μα. Νομίζω ότι δεν έχει καθόλου νόημα να μιλήσουμε πιο πολύ από 3-3,5 λεπτά. Και αν σωστά κατάλαβα, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πιο πολύ χρόνο στη διάθεσή τους και ξεπερνάνε και το χρόνο αυτό. Θα ήθελα να παρακαλέσω το εξής, να μην ε, ε, περιορίσουμε το χρόνο ομιλία. Αλλά αν γίνεται να τον γυρίσουμε σε δύο τμήματα, Γιατί άλλος κάποιο κάποιος 6,5-7 λεπτά και ε, δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Θα έλεγα λοιπόν να κόψουμε στη μέση, αν θέλει, το χρόνο ομιλία. Αυτό να έχει ο καθένα στη διάθεσή του 3-3,5 λεπτά κάθε φορά που μιλάει. Ερτούγκ, ne vous Κύριε Ερτούγκ, μην ανησυχείτε. Έχω τον κατάλογο εδώ μπροστά μου. Κανένα μέλο δεν πρόκειται να μιλήσει 5 ή 6 λεπτά έχει γίνει μία κατανομή έτσι ώστε να έχει 3,5 λεπτά ο καθένας maximum. Βεβαίως ε, ε, έχει γίνει μια κατανομη ετσι ωστε να εχει 35 λεπτα ο καθενας μάξιμου βεβαιως εχει γινει μια κατανομη του χρόνου αναλογική με βάση την δύναμη των πολιτικών ομάδων. Λοιπόν, ξεκινούμε το πρώτο πάνελ. Δεν έχετε τον κατάλογο, το σωστό κατάλογο παρεμβάσεων. Μην ανησυχείτε, εμπιστευτείτε την πρόεδρό σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις συζητήσεις με τον Ζεράρ Σίπερ από την Raw Control Route. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Θα το κάνω στα αγγλικά, γιατί έχω συνηθίσει να το κάνω στα αγγλικά την παρέμβασή μου. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σεβαστώ τα 7 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο μου δίνει την ευκαιρία να παρέμβω. Η Eurocontrol Route είναι μια οργάνωση για τη συνεργασία στον τομέα των οδικών μεταφορών που εδρεύει στο Μπενελούξ. Θα γίνει βεβαίω μια ανεξάρτητη αίτηση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Προ αυτή την κατεύθυνση Αφήνω λοιπόν το θέμα του Μπενελούξ. 15 μέλη ε, συμμετέχουν στην στον όμιλό μας, αναμένουμε και άλλα. Να δούμε λίγο τις διαφάνειες. Λοιπόν, θα είναι σύντομη αυτή η παρουσίαση, αφορά δύο ζητήματα. Την υπάρχουσα κατάσταση των οδικών μεταφορών και της εφαρμογής ε, της νομοθεσίας στην Ευρώπη και μία σκέψη σε ό,τι αφορά το πακέτο κινητικότητας. Όχι από πολιτικής πλευράς, αλλά από κοινωνικής πλευράς και κατά πόσο και από πλευράς αυτών που θα έχουν να εφαρμόσουν αυτή την νομοθεσία κυρίως. Λοιπόν, εάν δούμε την κατάσταση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των οδικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις εκθέσεις που λαμβάνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπουμε ότι έχουμε χάσει περίπου 80% των τρίτων εφαρμογής μετά την κρίση ε, του 2011. Ε, ε, έχουμε χάσει λοιπόν σημαντικό μέρος των ανθρωπίνων πόρων μας. Αν εξετάσουμε πιο προσεκτικά αυτά τα στοιχεία θα διαπιστώσετε ότι ε, αυτοί που είναι ε, καταρτισμένοι, εκπαιδευμένοι και μπορούν να εφαρμόσουν την νομοθεσία τότε θα χρειαζόμασταν 12 με 13 χιλιάδες ε, για, να, για τη σωστή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ 7 με 8 εκατομμύρια εμπορικά οχήματα, έτσι, για να καταλάβετε για τι μεγέθη μιλάμε. Να έχετε κατά νου επίσης ότι προτάσεις, στις προτάσεις αυτές υπάρχει μια διεύρυνση του πεδίου. Δεν αφορά πλέον μόνο τα φορτηγά. Στο προσεχές μέλλον θα συμπεριλαμβάνονται και τα πιο ελαφριά οχήματα, οπότε θα έχουμε ε, πολύ, περισσότερη δουλειά ακόμα στο μέλλον. Και θέλουμε βεβαίως ε, αυτή η εφαρμογή να ε, εφαρμόζεται με μια σωστή σχέση κόστος ωφέλους. Αν δείτε πώς συμβαίνουν αυτά σήμερα, ακολουθούμε λίγο την παλιά σχολή. με ιδέες δηλαδή εφαρμογής του 20ου αιώνα και όχι του 21ου αιώνα. Θα αναφερθώ επ' αυτού στη συνέχεια πρέπει να αντιμετωπίσουμε 20 με 30% απάτες σε ό,τι αφορά τους ταχυγράφους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εταιρείε μεταφορών ε, είναι ε, Οι περισσότερες εταιρείε είναι απολύτως νόμιμες και νομότυπες. Ε, υπάρχουν βεβαίως αυτό που θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να ονομάσει κανείς παραλιεύματα. Ε, είναι η ε, απάτη που έχει να κάνει με την εκπομπή και από εκεί πέρα έχουμε και τους ε, ε, οδηγούς που μεταφέρονται καθώς και τις, τις εταιρείε με εικονική έδρα είναι ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν επίσης από την πλευρά της εφαρμογής. Να δούμε τώρα λίγο το πακέτο για την κινητικότητα. Η νομοθεσία ε, σημαίνει ότι το 2019 θα αρχίσουμε να έχουμε τους ταχυγράφους. Θα υπάρξει όμως μια μακρά περίοδο εφαρμογής σε σχέση με την επικοινωνία μικρής εμβέλειας ε, εμείς πρέπει να εξετάσουμε εδώ ε, τις διάφορες γενιές ταχυγράφων και αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκο και θα περιπλακεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να το μελετήσουμε το θέμα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πακέτο κινητικότητας, εδώ υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ε, εβδομαδιαία ξεκούραση. Στο μέλλον θα διευκολυνθούν τα πράγματα. Ε, νομίζω ότι θα μπορέσει να εφαρμοθεί. Αν δούμε τι περιόδου αναφορά. θα πρέπει να δούμε και του ταχυγράφου σε σχέση με του ε, ψηφιακού ταχυγράφου που θα εφαρμοστούν σε σχέση με του συμβατικού. Ε, μιλάμε για ευελιξία ε, και η ευελιξία δεν πάει πάντα μαζί με την εφαρμοστικότητα. Πρέπει λοιπόν να, να ε, ενισχυθεί και η δυνατότητα εφαρμογή. Ορισμένε φορέ φαίνεται να μην είναι αρκετά ε, αυτά που συμβαίνουν και να, επίσης να παρεμβαίνουμε πολύ αργά. Εδώ υπάρχει μια καλή ιδέα, η οποία όμως δεν λύνει το πρόβλημα. Θέλουμε να έχουμε πραγματικές πληροφορίες για την εφαρμογή για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Και φτάνουμε τώρα ήδη στην τελευταία μου διαφάνεια, νομίζω πως δεν ξεπέρασα το χρόνο. Ε, κάποιες συστάσεις η εφαρμογή της καινοτομίας μέσω της τεχνολογίας. Έχουμε κάποια συστήματα, ε, το ANPR, η αναγνώριση των πινακίδων, ε, ηλεκτρονικά έγγραφα. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε όμως ότι πρέπει να έχουμε πρόσβαση να καταλάβουμε πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά 24 ώρες 24 ώρο, στις βάσεις δεδομένων και αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή ούτε καν στο ταχονέτ έχουμε πρόσβαση. Επίσης πρέπει να αναπτύξουμε πιο έξυπνες στρατηγικές εφαρμογής. Ε, εφαρμογή που να στην εμπιστοσύνη ή ε, ανταλλαγή δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο. Επίσης πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων που συμμετέχουν στις οδικές μεταφορές και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ιδανικά ε, μέσω της ε, ACR, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και ελπίζω ότι θα έχουμε μια καλή συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκύπερ. Και τώρα να δώσουμε τον λόγο στην επόμενη μελήτρα για τα λεπτά. Στην κυρία Μπερτελό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε εκπροσωπώ την ε, εθνική προσωπία των ε, Γάλλων ε, για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Είμαστε πάρα πολύ Ευρωπαίοι και θα επιμείνω σε αυτό. Συνεργαζόμαστε με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας πάντα σε ένα πνεύμα συμβαστικό και να σας πω ότι ήμασταν η πρώτη οργανώση του 2005 που απευθυνθήκαμε στο Ζακμπαρό, Επίτροπο των Μεταφορών, για να ρωτήσουμε κατά πόσον η απόσπαση ισχύει στο Καμποτάζ, γιατί από ό,τι φαίνεται κανείς δεν είχε θέσει την ερώτηση αυτή και πήρε πολύ καιρό μέχρι να έχουμε μία απάντηση και ακόμα η συζήτηση αυτή είναι σε εξέλιξη σήμερα. Η φιλοσοφία που ε, χαρακτηρίζει την οργάνωσή μας είναι η ρύθμιση, η οικονομική ρύθμιση για να βρούμε ίσους όρους ε, και για τα ελαφρά οχήματα και για να αποφύγουμε τον οδηματικό χαρακτήρα ζωής των ε, εργαζομένων. Θα ήθελα να σας δώσω λοιπόν κάποια στοιχεία μέσω που καταδεικνύουν την κατάσταση στην ευρωπαϊκή κατάσταση σε ό,τι αφορά τις γαλλικές επιχειρήσεις. Βλέπετε λοιπόν στο διάγραμμα αυτό μεταξύ στο 1993 στη γαλλική επικράτεια, ποια ήταν η εκπροσώπηση από γαλλικέ εταιρείε. Το 1993 ήταν 55,7%. Το 2016 είμαστε στο 10%. Αυτό τι σημαίνει ότι βασικά έχουμε διεθνεί διεθνείς μεταφορές στη γαλλική Επικράτεια πέρα από το transit, πέρα από την ε, απλή διέλευση. Δεύτερο γράφημα, δεύτερο διάγραμμα. Καταδεικνύει ότι το σύνολο των χιλιόμετρων σε διεθνείς μετάφορες πάντα στην γαλλική επικράτεια Από και προς τη Γαλλία δεν ε, γίνεται πλέον από γαλλικές επιχειρήσεις και μιλάμε για 6,9 δισεκατομμύρια των χιλιόμετρα σε ό,τι αφορά τα... τις διεθνείς δραστηριότητες των διεθνών επιχειρήσεων, θα προσέξετε ότι η Γαλλία το εθνικό επίπεδο μάλλον ε, των μεταφορών στην Γαλλία είναι 8%. Πριν από 20 χρόνια ήταν πολύ πιο υψηλό από ό,τι θυμάστε σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του καμποτάζου. Βλέπετε την κόκκινη γραμμή, ποιε είναι οι δραστηριότητε ε, ε, στην Γαλλία, οι μεταφορικέ δραστηριότητε για λογαριασμό τρίτων. Από το 1999 στο 2016 έχει μειωθεί κατά 15%. Ε, το καμποτάζ έχει πολλαπλασιαστεί κατά 5%. Κατά... Έχει πενταπλασιαστεί. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό το αγγίζει το καμποτάζ εδώ στο γράφημα βλέπετε τις ε, επτά μέσα σε διάστημα τριών ημερών όπως το 2009. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα ότι διεξεργάγεται μια πολύ δύσκολη ευρωπαϊκή συζήτηση για το γεγονός ότι οι Γάλλοι δεν είναι πλέον ε, ανταγωνιστική σε διεθνέ επίπεδο. Στο τελική ανάλυση αυτό δεν θεωρείται ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά γαλλικό πρόβλημα. Βρισκόμαστε λοιπόν πλέον σε μια ανοιχτή αγορά. Σε αυτή την ανοιχτή αγορά λοιπόν δεν έχουμε όλοι του ίδιου όρου, ούτε τι ίδιε αμοιβέ, ούτε και τι ίδιε κοινωνικέ εισφορέ. Βλέπετε λοιπόν εδώ στο διάγραμμα την κατανομή σε μπλε των κοινωνικών εισφορών και σε ό,τι αφορά την ε, αμοιβή των οδηγών και με κόκκινο το, κόστος μεταφοράς που δεν προσμετράται στην κοινωνική εισφορά. Δηλαδή δεν ε, ε, έχει να κάνει ούτε με τις εισφορές για την κοινωνική ασφάλεια, για τη συντάξη του καθεξής. Και βλέπετε στα δεξιά χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, μεγάλο είναι το τμήμα εκείνο το οποίο υπόκειται σε κοινωνικές εισφορές και βλέπετε στο αριστερό κομμάτι τι χώρε που δεν έχουν την ίδια αντιστοιχεία και αυτό προφανώ έχει να ε, επηρεάζει την δημοστικότητα. Ε, το πρώτο τελευταίο διάγραμμα, ώρε οδηγήσει οδηγήσεις σε στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Δεν θέλω να ξεκινήσω τις διαφωνίες, αλλά όταν βλέπουμε ότι είναι μεγάλη η διαφορά του κόστου οδήγησης των οδηγών κατά 80% τι εθνικό μέτρο να ληφθεί προκειμένου να αποκαταστήσει τους όρους ανταγωνισμού. Και στόχος της παρουσίασης αυτής και όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία είναι τα επίσημα στοιχεία της επίσημης Γαλλικής Αρχής και της Eurostat. Σκοπός λοιπόν είναι να καταδείξουμε ότι η συζήτηση την οποία κάνουμε σήμερα αντιμετωπίζουμε μια τεράστια δυσκολία. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε και το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε είναι ότι μια Ευρώπη τέτοια θα μας γυρίσει πίσω. Και βλέπουμε τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανώσεων, πάρα πολύ οξυμένες σε κάποια χώρα, κάποιες χώρες όπως και οι δικές μου, όπως και οι δικοί μου, κατηγορούνται για προστατευτισμό και κατηγορούνται για τις διάφορες θέσεις τους εναντί του πακέτου κινητικότητας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τους προτετασμούς, αλλά να κοιτάξουμε τα πράγματα και τα αριθμητικά στοιχεία όπως πραγματικά έχουν. Η πρόκληση είναι ότι οι στόχοι του πακέτου κινητικότητας είναι πολύ φιλόδοξοι. Με χαρά και συμμετέχουμε στην όλη διαδικασία και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κυρία Μπερτελό και όλοι δεν ξεπερνάτε το χρόνο ομιλία σας πάρα πολύ ωραία. Ο επόμενος ομιλητής. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Όλες οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα, είτε πρόκειται για το κοινωνικό πυλόν, είτε πρόκειται για την εσωτερική αγορά, ακόμα και όσον αφορά την απόσπαση, είναι όλες αλληλοεξαρτώμενες. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών, η ETF, έχει να κάνει συγκεκριμένε προτάσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, ατόμων και αγαθών, τηρώντας τους ευρωπαϊκούς κανόνες και κυρίως αυτό που είναι σημαντικό για την ETF είναι να μην υπάρχει καμία μισθολογική διακριτική μεταχείριση βάσει της εθνικότητος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πράξη βλέπουμε ότι το μέσο των δικών μεταφορών δεν είναι έτοιμος προκειμένου να ανοίξει εντελώς η σχετική αγορά. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει γράψει αυτό. Συνεπώς, το καμποτάζ πρέπει να παραμείνει μια προσωρινή δραστηριότητα. Ποιε είναι οι προτάσει τώρα τη Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών. Κάθε νέος κανονισμός, όπως και παλαιότεροι κανονισμοί. Θα πρέπει να έχουν ως στόχο να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου και επιβολή κυρώσεων εύκολα. Και θα πρέπει οι έλεγχοι να έχουν να κάνουν κυρίως με τον τοπισμό των παραβατών. Συνεπώς, ο ευφύης ταχογράφος με αυτόματο γεωγραφικό εντοπισμό του ECMR, τα εθνικά μητρώα, η πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους επιθεωρητές, είτε έχουν να κάνουν με τις μεταφορές είτε με την απασχόληση, καθώ επίση και τα εθνικά μητρώα οδικών μεταφορών είναι προτάσει που πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως και όχι το 2034. Όσον αφορά το καποντάζ θα πρέπει να έχουμε μόνο μία συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσα να πω τρει δραστηριότητες, γιατί κάνουμε ουσιαστικά διεθνή μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση. Η εκφόρτωση βέβαια αντιστοιχεί σε μία άλλη διεθνή μεταφορά. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέπετε μετά τη δραστηριότητα αυτή του καποντάζ μια περίοδο αναμονής 7 ημερών εκτός της επικράτειας καμποτάζ και θα πρέπει να προβλέπετε εκ των προτέρων μία δήλωση για κάθε μία τέτοια δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται σε συγκεκριμένο σημείο επαφή ευρωπαϊκό και το οποίο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Το όχημα θα πρέπει επίση να μπορεί να επιστρέφει τακτικά στην επιχειρησιακή του βάση. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε μόνο να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τι εικονικέ επιχειρήσει και τι επιχειρήσει γραμματοκιβωτίου, καταγράφοντα ουσιαστικά τη συγκεκριμένη αυτή δραστηριότητα του οχήματο στη χώρα που είναι καταγεγραμμένη και η επιχείρηση. Όσον αφορά την απόσπαση, οι κανόνε εδώ πέρα είναι σαφεί. Η οδηγία για την απόσπαση εφαρμόζεται στι δραστηριότητε του καποντάζ. Επ' αυτού δεν χωράει καμία αμφιβολία. Όσον αφορά τώρα τι διεθνεί μεταφορέ, η οδηγία για του αποσπασμένου εργαζομένου εφαρμόζεται μόνο όταν πληρούνται οι προποθέσει προβλέπονται στην οδηγία. Συνεπώ, το πρόβλημα για μα δεν έγκυται στου υφιστάμενου κανόνε, αλλά στην ελληπή εφαρμογή του ενδεχομένω. Όσον αφορά τώρα τον υφιστάμενο κανονισμό για το χρόνο οδήγηση και ανάπαυση, ο κανονισμός αυτός παρέχει αρκετή ευελιξία και η οργάνωσή μας, η ETF, δεν καταλαβαίνει τι άλλη ευελιξία ουσιαστικά θα πρέπει να παράσχουμε σε επιχειρήσεις. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του κανονισμού θα έχει επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των οδηγών, καθώς επίσης και στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς επίσης και στην ίδια την οδική ασφάλεια. Τώρα, το ζήτημα της επιστροφής στην έδρα, όπως αναφέρεται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώ ότι αποτελεί μια αυταπάτη. Στην πράξη, κανένα μέτρο δεν μπορεί να προστατεύσει τον πιο αδύναμο κρίκο, που είναι ουσιαστικά ο οδηγός και ο ίδιος ορισμός της έδρας είναι αρκετά σαφής. Και μην ξεχνάμε, όπως το έχει πει επανειλημμένος η ΙΤΕΦ, ότι όλα τα μέτρα αυτά είναι άλληλο εξαρτώμενα. Και αν μειώσουμε σε εβδομαδιαία βάση το χρόνο ανάπαυσης, τότε αυτόματα θα αυξήσουμε το χρόνο εργασίας και ορισμένοι κακόβουλοι μάλιστα θα θέλανε κατά αυτόν τον τρόπο να αυξήσουν και το χρόνο οδήγηση. Βλέπετε λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, στις 21 Νοεμβρίου η ΙΤΕΦ οργάνωσε πάρα πολλές διαδηλώσεις και δραστηριότητες παντού στην Ευρώπη και στα γαλλοβελγικά σύνορα. Διαδηλώσεις γιατί θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας προσέχει αρκετά ακόμα θεωρούμε ότι αν συνεχίσουμε να μην εισακόμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον, θα πρέπει να οργανώσουμε ακόμα πιο δυναμικέ διαδηλώσει. Αυτό που θέλουμε είναι να εφαρμόζονται και να τηρούνται οι φυστάμενοι κανόνε. Και κάθε νέο κανόνα θα πρέπει και αυτό με τη σειρά του να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο παντού. Όπω λένε άλλωστε και οι συνδικαλιστέ πολύ συχνά σε διάφορε χώρε, δεν συμφωνούμε για τίποτα μέχρι να συμφωνήσουμε για τα πάντα. Συνεπώς, αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε συνεχώς κατά νου είναι ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση η οποία είναι σίγουρα δυσχερής, αλλά που τελικά έχουμε δύο Ευρώπες και αυτό θα πρέπει να το λέμε. Από τη μία πλευρά έχουμε μια Ευρώπη που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες υφίσταται ένα πνεύμα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων και μια άλλη Ευρώπη όπου δεν υπάρχει καμία συλλογική σύμβαση, όπου οι οδηγοί πληρώνονται με μια απλή μερίσια αποζημίωση με βάση τα χιλιόμετρα που κάνουν και μάλιστα η πληρωμή τους αυτή είναι και εντελώ αδήλωτη. Θα θέλαμε λοιπόν πραγματικά να γίνει πραγματικό, πραγματικότητα αυτό που πάρα πολλέ φορέ έχει πει ο πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ, ότι δηλαδή για την ίδια εργασία θα πρέπει να προβλέπεται και η ίδια αμοιβή. Αυτό θα πρέπει να γίνει πράξη και να μην παραμείνουμε μόνο στα λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Λάσκο. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Φέρενσε Λάσκο, CEO της Βαμπρες International που είναι ένας παγκόσμιος παροχός υπηρεσιών και έχουμε τα αρχηγή του κεντρικού. γραφείο μας στην Ουγγαρία Έχουμε πάνω από 5.000 ε, επαγγελματίε οδηγούς στην εταιρεία μας και θα ήθελα να σας δώσω κάποιες ε, ρεαλιστικές πτυχές αυτού του πακέτου κινητικότητας. Εμείς δεν είμαι πολιτικός, είμαι απλά ε, μια εταιρεία ε, μεταφορών. Είμαστε λοιπόν καταχωρισμένοι στο χρηματιστήριο της Βουδαπέστης, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι λοιπόν είμαστε απόλυτα διαφανεί στον τομέα των μεταφορών. Συνάδουμε και συμβαδίζουμε με όλες τις ευρωπαϊκές διατάξει όπως κάθε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποιες πτυχές του ζητήματος και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δυστυχώς ε, είχαμε καταλάβει άξιο καταλαβαίνουμε η συζήτηση και η διαβούλευση πριν από το πακέτο κινητικότητα δεν ήταν αρκετά ευρεία και ει βάθος και έτσι οι κατασκευαστέ και οι καταναλωτές θα έπρεπε να είχαν εκφράσει και αυτή μια γνώμη γιατί όλοι εξ αυτών θα επηρεαστούν από το πακέτο κινητικότητα. Θα ήθελα να σας καταδείξω λοιπόν τη σημασία του τομέα των οδικών μεταφορών στην Ευρώπη. 75% των ε, παρόχων, ε, μάλλον των μεταφορών, γίνεται μέσω των δρόμων. Και περίπου 71% του ΑΕΠ των ε, μεταφορών έρχεται από τον τομέα των οδικών μεταφορών στην Βουλγαρία και στην Ισπανία είναι 13%. 65% κατά μέσο όρο γίνονται οι, οδικές μεταφορές, οι μεταφορές μέσω οδικών οδηγών. 80% των εθνικών μεταφορών που γίνεται από την Ευρώπη των 15, τα παλιά κράτη-μέλη, και μόνο 20% από τα καινούργια κράτη-μέλη. Το διεθνές σκέλος, η αναλογία είναι αντίθετη σχεδόν, αντίστροφη. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν είναι αυτή η ε, ανακατανομή ε, των ε, κρατών μελών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει. Οι κανόνες των μεταφορών είναι σωστοί σήμερα. Γιατί? Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κλάδο θα μπορούσε να οργανώνεται με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι σήμερα, αλλά υπάρχουν και κάποιε συνέπειε. Για παράδειγμα, αύξηση των τιμών κατά 30%, 20% και αυτό θα φανεί στην ε, τελική τιμή του προϊόντος. Μια αισθητή, ένας αισθητός πληθωρισμός και επίσης μπορεί να τραχτεί και η αλυσίδα παροχής των προϊόντων, αν επαρκώς ε, υπόψη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και τέλος, αυτή η αύξηση του κόστους μεταφοράς θα μπορούσε να μειώσει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Δεν θέλω όμως να μιλήσω για τα μακροοικονομικά ζητήματα, να δούμε το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης το πακέτο κινητικότητα δεν εξυπηρετεί τα κοινωνικά συμφέροντα των οδηγών, γιατί δεν έχουμε αρκετού ε, στου δρόμου για να. Και αυτά που προβλέπονται δεν είναι άνετα για τους οδηγούς. Αν λοιπόν οι οδηγοί αφήσουν ε, τα φορτηγά τους ε, αφύλακτα στους αυτοκινητοδρόμους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για αυτούς από λόγω της μετανάστευσης και λόγω άλλων ε, υποθέσεων. Ο Επίτροπος επίσης ε, επισκέφθηκε την Ουγγαρία και παραδέχτηκε ότι η έλλειψη χώρων στάθμευσης και ξενοδοχείων αποτελεί πραγματικό ζήτημα και άρα δεν ε, είναι εφικτό αυτό που προβλέπετε για τον τομέα των μεταφορών. Άρα προτείνουμε να υπάρξει ένας κανονισμός όχι για τρεις εβδομάδες, αλλά για τέσσερις εβδομάδες σε ό,τι αφορά το μέγιστο όριο που μπορεί κανείς να μείνει στο δρόμο και μετά από τις τέσσερις αυτές ημέρες να μπορεί να πάει κανείς τρεις-τέσσερις ημέρες στο σπίτι του με την οικογένειά του. Αυτό είναι προς το κοινωνικό συμφέρον του οδηγού. Και ως Ουγγρική εταιρεία θα σας προκαλέσει εντύπωση ότι υποστηρίζουμε αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε για παράδειγμα την οδηγία για την απόσπαση. Θα καλωσορίζαμε μια τέτοια ρύθμιση και οι 5.000 οδηγοί μας σε κάθε περίπτωση για να προωθήσουμε τον δίκαιο ανταγωνισμό και την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία στην Ευρώπη. Ωστόσο, η πρόταση αυτή, όπως έχει σήμερα, δεν επιτρέπει τις ε, διεθνείς μεταφορές. Φανταστείτε. Φανταστείτε έναν ε, οδηγό σε ένα διεθνέ ε, ταξίδι. Να αλλάζει χώρα κάθε μια-δύο μέρες. Ε, και αυτή, αυτός ο οδηγός λοιπόν και αυτή η εταιρεία θα πρέπει να πληρεί τους εκάστοτε όρους της κάθε χώρας. Διαφορετική νομική ομορφία της διατάξης, διαφορετική εκπρόσωπη του νόμου, διαφορετική γλώσσα. Θα πρέπει να υπάρχει μια δυο μέρε. και αυτη αυτος ο οδηγο λοιπον και αυτη η εταιρεια θα πρεπει να πληρει του εκαστοτε ορου τη καθε σε διαφορετικη νομικη ομιλια τη διαταξης διαφορετικη εκπροσωπη του νομου διαφορετικη γλωσσα θα πρεπει να υπαρχει μια ενιαια καταχωρηση αυτό το τεχνικό θα ήταν απόλυτα δυνατόν. Πρότασή μας λοιπόν θα ήταν ε, για 10 ημέρες ε, ανάχωρα αναμήνα απορρίθμιση και πιστεύω ότι αυτό κλείνει όλα τα κενά. Αυτό θα καταπολεμούσε τον αθέμητο ανταγωνισμό, το κοινωνικό dumping. Θα, επιτρέπε, θα επέτρεπε όμως τη σωστή αποτελεσματική λύση του διεθνού σκέλου των μεταφορών. Αγαπητοί βουλευτέ. η απόφαση προφανώ στα χέρια σα βρίσκεται να μην ξεχάσετε ότι το πακέτο κινητικότητα θα έχει πολύ πιο πολλέ επιπτώσει πέρα από τη ρυθμίση του κλάδου. Έχει σοβαρέ συνέπειε για το ευρωπαϊκό ΑΕΠ, την ανταγωνιστικότητα και τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Ευχαριστώ πολύ. Εμεί ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση σε αυτή. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Πολόνιο, για 7 λεπτά παρακαλώ έχετε το λόγο. Ανοίξτε όμως το μικρόφωνο σας παρακαλώ πρώτα. Λοιπόν, μηδενίζω πάλι το χρόνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εκπροσωπώ την Άντραμα, Εθνική Ένωση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών που υφίσταται από τη δεκαετία του 50 στην Πορτογαλία. Με συγχωρείτε, δεκαετία του 70, από το 1975. Συμμετέχουν στην Ένωση αυτή χιλιάδες ε, επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που έχουν συνολικά 35.000 ε, φορτηγά και ασχολούνται όχι μόνο με χώρες αλλά και με διεθνείς εμπορικές μεταφορές. Όσον αφορά τώρα τον ορισμό της απόσπασης εργαζομένων, όπως προβλέπεται σχετική οδηγία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν υπάρχουν ε, τροποποιήσεις όσον αφορά το πρώτο άρθρο της οδηγίας του 1996 και επίσης ε, στο δεύτερο άρθρο δεν βλέπουμε να υπάρχουν αλλαγές. Δηλαδή παραμένει σαφές τα δύο αυτά άρθρα ότι ε, απόσπαση μπορούμε να έχουμε σε συγκεκριμένου μόνους τομείς και όχι στον τομέα των μεταφορών. Και εφόσον προβλέπεται στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει αυτό να γίνεται στα πλαίσια μιας σύμβασης μεταξύ δύο μόνο κρατών και όχι μεταξύ πολλών διαφορετικών κρατών. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τον τομέα των μεταφορών, εμεί είμαστε ένα κλάδο όπου έχουμε πολλέ διαφορετικέ δραστηριότητε οι οποίε εκτελήσονται παράλληλα και ξέρετε ότι οι περισσότεροι οδηγοί τελικά διασχίζουν όχι μόνο μία και δύο, αλλά πάνω από δύο χώρες. Αυτό ουσιαστικά αντιτίθεται στα όσα λέει η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Ένα οδηγό ο οποίο επιτελεί διεθνεί οδικέ εμπορευματικέ μεταφορέ δουλεύει εκτό τη χώρα του και πολλέ φορέ, όπω σα είπα, χρειάζεται να περάσει από πολλέ διαφορετικέ χώρε. Αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εξαίρεση και παρέκκληση. Αυτή είναι, αν θέλετε, η πιο συνήθι φύση εργασίας ενός οδηγού. Μέχρι στιγμή δεν καλύπτονται οι περιπτώσει αυτέ από την οδηγία απόσπαση εργαζομένων. Όταν λέμε επίση ότι πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη σύμβαση, α πούμε, ότι ένα οδηγό φεύγει από την Πορτογαλία για να πάει στη Γαλλία και α πούμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη σύμβαση με ένα πελάτη. Αν εγκαταλείψει εν συνεχή ο οδηγό αυτό στην Γαλλία και πάει σε μια άλλη χώρα, θα πρέπει να προβλεφθούν και άλλε τέτοιε συμβάσει για να καλύψουν την εργασία του. Α δούμε πείτε τώρα τον κανονισμό 1072 του 2009 που δίνεται ένα ορισμό όσον αφορά τι διεθνεί ε, εμπορικέ μεταφορέ. Πάλι δεν θεωρώ ότι όσα προβλέπετε εδώ πέρα θα μπορούσαν να ενταχθούν στα πλαίσια τη οδηγία απόσπαση εργαζομένων εφόσον δεν υπάρχει ακόμα το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο. Οι ε, υφιστάμενε προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροποποίηση οδηγία αυτή δεν καλύπτουν και τι περιπτώσει εκείνε τι οποίε σα ανέφερα. Όπως σας είπα, στον τομέα των μεταφορών έχουμε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε όχι μόνο Πορτογάλους οδηγούς, αλλά οδηγούς, για παράδειγμα, από την Ουγγαρία, όπως ανέφερε πριν από λίγο ο μιλητής από την Ουγγαρία. Και ε, εκεί πέρα μπορεί τελικά να προκύψουν ε, πολλέ διαφορετικέ μορφέ εργασία. Ενδεχομένω ο άνθρωπο αυτό ξεκινώντα από την Ουγγαρία να πρέπει να κάνει 5, 6, 7 διαφορετικέ παραδόσει σε διάφορε χώρε και θα πρέπει επίση ε, ο οδηγό αυτό από την Ουγγαρία, εφόσον για παράδειγμα δραστηριοποιείται στη Γαλλία, να λαμβάνει και μία επιπλέον αποζημίωση, καθότι εκεί πέρα το βιωτικό επίπεδο είναι πιο υψηλό και η ζωή πιο ακριβή. Ξέρετε ότι ε, πολλέ φορέ οι οδηγοί εργάζονται μόνοι τους, δεν χρειάζεται κάθε φορά να φέρουν μαζί και την οικογένειά τους και κατά αυτόν τον τρόπο διαφέρουν ουσιαστικά από τους υπόλοιπους αποσπασμένους εργαζομένους. Εμείς δεν είμαστε μία από τις πιο κεντρικές ή οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, δεν θα είχαμε ενδεχομένω το πιο υψηλό κόστος ή τις πιο υψηλές αμοιβέ. Αν δείτε για παράδειγμα όντως το κόστος για τη Γαλλία όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, σίγουρα το κόστο του είναι πάρα πολύ ψηλό και εξαιτία του διεθνού ανταγωνισμού ενδεχομένω να χάνουν όλο και περισσότερο μερίδιο τη αγορά. Αυτό ισχύει για διάφορε προηγμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω η Γαλλία. Όμω το ζήτημα αυτό πάλι δεν μπορεί να διευθετηθεί από μόνο του από την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Α δούμε μια άλλη πτυχή τώρα του προβλήματο. Συνεργαζόμαστε με διάφορες άλλες ενώσεις και συλλόγους και από κοινού προσπαθούμε να μην δώσουμε την υποστήριξή μας, θα αποφασίζεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθότι η δραστηριότητά μας είναι πολύ σχηδής και διαφέρει πάρα πολύ από την μία επιχείρηση στην άλλη. Μεγάλες αλλαγές παρατηρούνται, μεγάλες διαφορές με συγχωρείτε παρατηρούνται και από τη μία χώρα στην άλλη, για παράδειγμα ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Υπάρχουν πολλά φόρα πάντως που ασχολούνται με την αυτή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων. Ξέρετε ότι μερικές επιχειρήσεις απαιτούν από τους οδηγούς να επιστρέψουν στην έδρα τους μετά από μία ή περισσότερες εβδομάδες εργασίας. Να δείτε τώρα πώς έχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε την ε, τακτική εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης εντός και εκτός καμπίνας. Το πρόβλημα είναι πώς μπορεί να καταγράψει κανείς και τη, τα Σαββατοκύριακα. Ξέρετε ότι ε, ε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πετύσουμε από τους οδηγούς να συμμορφωθούν εντελώς με τον κανονισμό αυτό όταν αυτό δεν συνάδει καθόλου με την φύση του επαγγελματό τους. Όταν επιβάλλουμε μία δεκάλεπτη ανάπαυση του οδηγού στην καμπίνα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο από όλους τους οδηγούς, γιατί εξαρτάται πάρα πολύ από το επαγγελματικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν. Βλέπετε στον πίνακα αυτό κάποια αριθμητικά δεδομένα που θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου Στον πίνακα αυτού η Πορτογαλία βρίσκεται όπως βλέπετε στην 11η θέση και ένα 66% των οδικών μεταφορών μας, των εμπορικών, είναι διεθνείς. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα επίσης των διεθνών οδικών μεταφορών που λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία εκτελούνται από Πορτογάλους οδηγούς. Ας πάρουμε και τη Γερμανία. Βλέπετε ότι Έχουμε εδώ πέρα πολύ σημαντικούς οικονομικούς κλάδους στη χώρα αυτή που εξυπηρετούνται και αυτοί με τη σειρά τους από Πορτογάλους οδηγούς όσον αφορά πάλι το τμήμα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Πέρα από τους κανόνες που ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε και κανόνες οι οποίοι ισχύουν προφανώς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες πολλές φορές δημιουργούν ένα πιο έντονο ανταγωνισμό μεταξύ ημών Ευρωπαίων οδηγών και οδηγών από τρίτες χώρες. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση ιδιαίτερα χαοτική, αν δεν υπάρξει τελικά εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων. Ο Βίλατσεν το λόγο. Øh, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι παρουσιάσει και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για το γεγονό ότι έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη θέση μα. Είμαι πρόεδρο τη 3F Transport, αλλά και για την εταιρεία σκανδιναβικών μεταφορών. Ήμουν και εγώ οδηγό στην δεκαετία του 80 και του 90 μετέφερα από την Δανία προς την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, ψάρια και άλλα τρόφιμα. Ήταν καλή δουλειά με μια ελευθερία, με μια σωστή αμοιβή, με φίλους και φιλίες σε όλες τις χώρες. Σας ε, μοίρασα και την έκθεση αυτή η οποία καταρτίστηκε από την 3F Transport σε συνεργασία με τους Δανούς εργαζοντές. Πρόκειται για μια διαδικασία α, και για εταιρείε οι οποίε έχουν α, ε, οδηγοί οι οποίοι 7 εβδομάδε ε, ζουν μέσα στα φορτηγά του και βγάζουν μόνο το 1 τρίτο του μισθού από αυτά που βγάζουν οι Δανείοι, οι Μακεδόνε στην και πιστεύω ότι είναι σημαντική λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά και είναι σημαντικό το θέμα τη ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών. Αλλά ο στόχο αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται ει βάρο εις ε, ε, ίσων όρων αμοιβή και διαβίωση για του Ευρωπαίου πολίτε. Δεν μπορεί να είναι αυτό αποδεκτό. Βάσει δηλαδή αθέμη του ανταγωνισμού να συμβαίνουν όλα αυτά. Και ξέρω ότι πιο πολύ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν με την αρχή αυτή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλωστε. Γι' αυτό και είμαι θετικό. Έχω θετική, ε, είμαι θετικά διακείμενο προ το πακέτο κινητικότητα ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα κάτι συγκεκριμένο για τι προτάσει, για την ε, απόσπαση. Συμφωνούμε, συμφωνούμε στην πρόταση αυτή να αναγνωρίσει ότι ε, ο κάθε οδηγό είναι αποσπασμένο ουσιαστικά σε άλλη χώρα όταν δουλεύει σε άλλη χώρα και θα πρέπει να αποζημιώνεται σύμφωνα με του όρου που επικρατούν στη χώρα που δουλεύει. Αυτό είναι απαραίτητο. Και ο τομέα των μεταφορών προφανώ πρέπει να έχει ειδική ρυθμίση σε ό,τι αφορά την οδηγία για την απόσπιση οριοτριών ημερών, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να βγάζουν νόημα ε, να μετράτε δηλαδή τρεις ημέρες μετά από την απομάκρυνση από τη χώρα του, όχι σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Καταλαβαίνω φυσικά το επιχείρημα ότι θα υπάρχει πολυγραφειοκρατία, γραφειοκρατία, αλλά πολύ απλά θα πρέπει να επιληθεί το ζήτημα. Θα, πρέ... θα μπορούσαμε να συζητήσουμε άλλα μοντέλα που επιτυχάνουν το ίδιο στόχο. Για παράδειγμα, η διεθνεί ε, οδηγοί να αποζημιώνονται σύμφωνα με τους όρους της χώρας στην οποία μεταφέρουν τα αγαθά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το καμποτάζ, συμφωνούμε και την καλωσορίζουμε. Πρόκειται για διεθνείς μεταφορές, οι οποίες θα πρέπει να την χάνουν αποζημίωση σύμφωνα με την χώρα στην οποία γίνεται η μεταφορά. Από την πρώτη μέρα, αν αποφασιστεί αυτό, τότε θα μπορέσει και η Ένωση μας να υποστηρίξει την απεριόριστη οδήγηση σε πλαίσιο πέντε ημερών και σε ό,τι αφορά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι συνδυαζόμενε μεταφορέ, είμαστε λίγο έκπληκτοι γιατί κινείται προ την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν θέλουμε να υπάρχουν αντίθετοι κανόνε σε ό,τι αφορά την αποζημίωση και του ε, συνθήκε εργασία. Θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι οι συγκεκριμένοι κανόνε, μάλλον οι υφιστάμενοι κανόνε για την χρόνο οδήγηση και αναπαυση θα πρέπει να τηρηθούν. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τι ώρε ανάπαυση κτλ. Και θα μπορεί να ισχύει και ένας προσωρινός ε, χώρος ανάπαυση δεν χρειάζεται να είναι το σπίτι. Γιατί φυσικά οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν και τα προϊόντα του. Και άρα δεν είναι σωστή η ισορροπία να προτείνουμε 20 συναπτέ ημέρε. Χρειαζόμαστε λοιπόν και ε, ξεκούραστους οδηγού. Αυτές είναι οι τρεις νέες προτάσεις ε, σε ό,τι αφορά τους οδηγούς. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει και επιτήρηση, γιατί δεν έχει νόημα να υπάρχουν οι κανόνες αν δεν υπάρχει επιτήρηση. Και υπάρχουν τρία εργαλεία. Η σύγχρονη ταχογράφη καταρχάς για ψηφιακή, ψηφιακό έλεγχο και ψηφιακές ε, συμβάσεις, ψηφιακή αποζημίωση και ψηφιακή αποθήκευση όλων των δεδομένων της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ε, ασφάλειας και οποιασδήποτε άλλη ασφάλεια και επίσης ε, ψηφιακή καταχώρηση των, ε, της, των συνόρων που περνάει κανείς και του τρόπου οδήγηση και γνωρίζουμε από το GPS πως ε, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αυτές. Αν μπορούμε λοιπόν να συνδυάσουμε αυτές τις δύο τεχνολογίες, μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά ε, ψηφιακά και έτσι μπορούν οι αρχές να διεξαγάγουν πιο αποτελεσματικούς ε, ε ελέγχους. Δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς δηλαδή το 2030 και ούτω καθεξής για να εισαγάγει ψηφιακούς ταχογράφους. Όχι, μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά τώρα. Δεύτερη, δεύτερο εργαλείο που πρότεινε και ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εργασίας. Ε, αυτό ε, εξάγγειλε στην ε, δήλωση για την κατάσταση της Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή συνεργασία, ευρωπαϊκό συντονισμό σε ό,τι αφορά την δίκαιο ανταγωνισμό και τον σωστούς όρους για τους υπαλλήλους, για τους οδηγούς. Θα πρέπει να υπάρχουν σωστά στατιστικά στοιχεία και για την οδηγούς και για το χρόνο εργασία. Ευρωπαϊκή Αρχή λοιπόν εργασία, εξαιρετικό εργαλείο θα μπορούσε να αποτελέσει αυτό για την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, διάφορα μέτρα και θα πρέπει να συνεργαστούμε αν θέλουμε καλέ συνθήκε εργασία. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία και με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή Μεταφορών και αυτό προ το συμφέρον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των ευρωπαϊκών οδηγών και τη συνοχή τη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο καθηγητής Μπορκόφσκι έχει το λόγο από το Πανεπιστήμιο του Γκτάνσκ. Yes, I Εκπροσωπώ το Πανεπιστήμιο του Γκτάνσκ που έχει μεγάλη εμπειρία έρευνα στον τομέα των μεταφορών. Έχουμε προετοιμάσει λοιπόν εδώ μια παρουσίαση με κάποια αποτελέσματα στα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα. Έχουμε περίπου 20 με 30 χρόνια εμπειρία σε ό,τι αφορά την έρευνα στον τομέα των μεταφορών. Λοιπόν, υπάρχουν δύο μελέτες Η μία αφορά τις εταιρείε μεταφορών ε, στην Πολωνία και τον επίπτωση για το πακέτο κινητικότητας. Βεβαίως μπορεί να μην πολύ η Πολωνία, αλλά αυτά που αναφέρονται εδώ αφορούν όλες τις χώρες της Ένωσης και αφορά ε, και τις περιφερειακές χώρες της Ένωσης. Ε, θα δείτε στη συνέχεια την ευρύτερη εικόνα, τη δεύτερη μελέτη δηλαδή, τη σχέση μεταξύ την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών και την ε, γενικότερη οικονομική ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Λοιπόν, ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, στα έσοδα ε, και στις επιχειρήσεις. Εδώ έχουμε το καμποτάζ που περιορίζεται στις πέντε μέρες, την απαγόρευση στην, την, να κοιμάται κάποιος τα οχήματα και την ε, απόσπαση που θα εφαρμόζεται μετά από πέντε μέρες. Ε, πήγαμε ως το τέρμα, παρότι είχαν αλλάξει έκτοτε κάποια πράγματα ε, στην νομοθεσία, αλλά επειδή είχε αρχίσει η μελέτη δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε κάτι από εκεί πέρα. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τα αποτελέσματα, η μείωση στον αριθμό των, ε, της δραστηριότητα ε, για πάνω από 7% αφορά τα 2 τρίτα ε, των ε, εταιριών. Τώρα για τα έσοδα. Η μείωση είναι για πάνω από 5% και τουλάχιστον 50% ε, των επιχειρήσεων, ίσως και περισσότερες. Για όσους γνωρίζουν καλά τον τομέα των μεταφορών, θα ξέρετε ότι οι περισσότερες εταιρείε ε, έχουν πολύ ε, λίγα περιθώρια κέρδους. Οπότε 5% μείωση εσόδων σημαίνει πτώχευση, έτσι. Βεβαίω μπορεί αυτό να αντισταθμιστεί με τη μείωση του κόστου. Όμω ε, δυστυχώ μείωση του κόστου δεν μπορεί να υπάρξει. Θα έχουμε αύξηση τουλάχιστον 5% για τουλάχιστον 5% των επιχειρήσεων και αυτή η αύξηση θα είναι κυρίως ορατή στο εργατικό κόστος όπου μπορεί να έχουμε έω και 50-60% ε, αύξηση ιδιαίτερα με την νομοθεσία περί απόσπασης. Λοιπόν, πώς αυτό μεταφράζεται τώρα στο τι συμβαίνει ε, στις διάφορες εταιρείε. Οι εταιρείε θα πρέπει προφανώς να μειώσουν ε, το στόλο τους. Γιατί, γιατί πρέπει να πληρώσουν ε, για, την, για το δάνειό τους ή για την ενοικίαση και δεν θα μπορούν βεβαίως να πληρώσουν τις δόσεις τους και τα επιτόκια. Η μείωση για τις μικρές επιχειρήσεις πάνω από 50% ε, αφορά περίπου όλες τις εταιρείες, 90%. Ε, εάν λοιπόν έχουμε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση με δύο φορτίγα, ε, ουσιαστικά είναι σαν να την αποσύρουμε από την αγορά. Από εκεί πέρα έχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις όπου η μείωση είναι λιγότερο σημαντική, αλλά και πάλι είμαστε κοντά στο 50%. 50% των επιχειρήσεων λέει δηλαδή, θα χάσουν 10% των οχημάτων. Τώρα για την απασχόληση. 90% των επιχειρήσεων στις μικρές επιχειρήσεις ε, αναμένουν, αναμένεται να απολύσουν 30% του προσωπικού τους. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι, μιλάμε για αυτές δηλαδή που έχουν 1 έως 9 εργαζόμενους. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις εκεί πέρα βεβαίως υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ε, ε, προσαρμογής, οπότε το σοκ θα είναι λιγότερο ισχυρό η μείωση θα είναι της τάξης του 20% θα και θα αφορά 30% των επιχειρήσεων. Και τέλος ε, έχουμε τα, ε, τα άδεια φορτηγά. Εάν προσθέσουμε τη νομοθεσία περί απόσπασης ε, δεν υπάρχει δυνατότητα ξεκούρασης μέσα στο αυτοκίνητο, θα αυξηθούν κατά 7% τουλάχιστον οι μεταφορές με άδειο φορτίο. και βεβαίως η επίπτωση είναι το περιβαλλοντικό ε, η περιβαλλοντική ζημία, θα έχουμε περισσότερη βενζίνη, περισσότερες εκπομπές. Θα δούμε τώρα την ευρύτερη εικόνα. Προσπαθήσαμε να συνδέσουμε το ΑΕΠ με διάφορους δείκτες για την απόδοση του τομέα των μεταφορών. Στην πρώτη στήλη βλέπετε τη σχέση ε, του σωματικών μεταφορών στον τομέα τη απασχόληση, εδώ είναι λίγο πολύ ίδια τα πράγματα σε όλε τι χώρε. Όμω είναι πολύ πιο ισχυρό, ισχυρή η διαφορά για τι χώρε τη περιφέρεια σε σχέση με τι χώρε του πυρήνα. Αυτό σημαίνει ότι η ρυθμή ανάπτυξη στο ΑΕΠ στι περιφερειακέ χώρε εξαρτάται περισσότερο από τι μεταφορέ από ό,τι στι ε, χώρε του πυρήνα, του κέντρου. Εάν δείτε τώρα τη δεύτερη στήλη, εδώ βλέπουμε τον αριθμό των επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών που δεν αυξήθηκε απαραίτητα για κάποιες χώρες παρότι υπήρξε αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες χώρες υπάρχει μια πλειοψηφία μεγάλων επιχειρήσεων που ε, δεσπόζουν στην αγορά και σε άλλες χώρες έχουμε πιο πολλές μικρές επιχειρήσεις. Στις δύο επόμενες στήλε διαπιστώνουμε ότι οι χώρες του πυρήνα η απόδοσή τους ε, ε, στον τομέα των μεταφορών ε, βασίζεται κυρίως στο κεφάλαιο ενώ οι περιφερειακές χώρες περισσότερο στην εργατικό δυναμικό. Λοιπόν, συνοψίζοντας, οι οδικές μεταφορές στην Ευρώπη αποτελείται από μικρές επιχειρήσεις ενώ για την Ευρώπη των 15 είναι κυρίως οι μεγάλες, είναι κυρίως μεγάλες εταιρείες. Βεβαίω οι μικρέ επιχειρήσει ε, είναι πιο δύσκολο να προσαρμοστούν στο σοκ ε, τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ιδίω από τη στιγμή που αυτή η πρόταση αφορά μόνο ένα σκέλος της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή την, την εργασία. Αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο επίπεδο κεφαλαίων. Μπορεί εύκολα δηλαδή να ε, βρουν, να μοχλεύσουν κεφάλαια. Τώρα, οι επιπτώσεις, οι παρενέργειες, λιγότερο ανταγωνιστική αγορά, λιγότερη ρυθμία, μικρότερη ρυθμία ανάπτυξη, ιδιαίτερα στι περιφερειακέ χώρε, όλε τι περιφερειακέ χώρε. Όχι μόνο δηλαδή τι χώρε τη διεύρυνση, αλλά και τη Ευρώπη των 15. Αυτά ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρίε και κύριοι εμπειρογνώμονε, σα ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο. Τώρα θα γίνει η συζήτηση. Πώς θα γίνει αυτή η συζήτηση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έχετε αυτό το χαρτί με τον χρόνο ομιλίας και έχετε τρία λεπτά μας χάρη ναι, εσείς κύριε Βαντενκάμπ για να ε, διαλέξετε σε ποιον απευθύνεστε και να υπάρξει απάντηση. Κύριε Βαντενκόπ, τρέχει ο χρόνος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τρεις ερωτήσει να κάνω προς τον κύριο Σχίπερ και σε ό,τι αφορά... Α, μάλλον θα ήθελα να μου τις απαντήσει με ένα ναι και με ένα όχι, γιατί μιλάμε για πινκ-πονγκ. Ε, θα πρέπει με συντομία να απαντήσει. Καταρχάς, ε, μπορούμε να κτιτηρήσουμε όλες τις κοινωνικές παροχέ ε, παροχές μέσω του ηλεκτρονικού ταχογράφου και γιατί όχι. Τι εννοείται, όλες τις κοινωνικές προβλέψεις, του χρόνου ανάπαυσης, καμποτάζ, ε, σύνορα κτλ. Έτσι, ναι, θα μπορούσαμε. Αν το φέρετε έτσι, θα μπορούσαμε, ναι. Θα μπορούσαμε να τους εισαγάγουμε από το 2022. Από μένα, από δική μου πλευρά, ναι, Σαφέ και αυτό. Λέει ναι, μου. Και η περίοδο αναφορά θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο πίσω από 28 ημέρες, πιο πολύ 28 ημέρες. Αν θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε αυτό τεχνικά, ε, θα μπορούσαμε. Ε, αλλά δεν έχω απάντηση. Θα θέλετε να μου το πείτε, να το κοιτάξετε και να μου το πείτε. Μάλιστα, να περάσω στον κύριο από τα τώρα. Τον κύριο Παρίλιο. Αυτό το σχέδιο μπορεί να γίνει πραγματικότητα χωρίς επιπλέον ξενοδοχεία. Αυτή είναι η ερώτηση των 5 ευρώ. Ακούστε, το πρόβλημα δεν είναι τα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα είναι η υποστήριξη που έχουν οι επιχειρήσεις, η λογιστική υποστήριξη. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς τον κύριο Βάμπεριχ. Έχετε περάσει στις 28 ημέρες ποτέ στο... στην καμπίνα του φορτηγού. Ναι. Πώς σας φάνηκε. Είναι διαφορετική δουλειά. Αλλά πιστεύω ότι ένας οδηγός ε, μπορεί να κάνει πέντε φορές ε, παραπάνω. Ε, να βγάλει πέντε φορές τον ουγγρικό κατά το μισθό, οπότε έχει διαφορά. Προς τον κύριο Πρωτοβουλία, λέει ο κ. Φοντεγκάμπ, μια ερώτηση να κάνω. Ακούστε, εγώ, ο πατέρας μου, ο παππούς μου, είμαστε όλοι οδηγοί, όλη μας τη ζωή. Είμαστε στο τομέα μεταφορών τόσα χρόνια και ξέρω ακριβώς τι σημαίνει να είναι κάποιος σε ένα φορτηγό και να κοιμάται εκεί. 28 μέρες μέσα στο φορτηγό ε, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα που να είσαι εδώ 8 μέρες 8 ε, ώρες τη μέρα. Μια ερώτηση για τον καθηγητή από το Gdansk. Ε, όχι, τα τρία λεπτά τα περάσατε. Ο κύριος Νίλσον έχει το λόγο τώρα. Για τρία λεπτά πινκ-πονγκ. Ευχαριστώ. Uh, Δύο ερωτήσει έχω να κάνω προς τον κύριο Λάικο. Πρώτη ερώτηση. Η εξή. Πόσο μεγάλο ποσοστό των ε, αποστάσεων που κάνετε είναι πραγματικές αποστάσεις καμποτάζ. 0%. Eh, eh, Κάτι τώρα, μια άλλη ερώτηση που θα ε, προαπαιτήσει ίσως μια πιο εκτεταμένη απάντηση. Αν ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πακέτο κινητικότητας περάσει, δεν θα το αλλάξουμε στο Κοινοβούλιο. Αν συνέβαινε αυτό, τι αλλαγέ θα έπρεπε να κάνετε στην επιχείρησή σα, για να εξακολουθήσετε να ενεργείτε και να λειτουργείτε στην διεθνή αγορά μεταφορών. Τι, απαιτεί, αλλαγές θα απαιτούσε λοιπόν η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την επιχείρησή σα. So, την παρουσίασή μου, είπα ποια είναι τα σημεία κλειδιά όπου θεωρούμε ότι πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν και να είναι διαφορετικά. Δύο είναι κυρίως τα σημεία. Οι 45 ώρες στην καμπίνα, τέσσερις εβδομάδες maximum, ε, χωρίς να πηγαίνει σε ένα κέντρο ξεκούρασης οδηγών, αλλά να γυρίζει σπίτι του, είναι καλύτερο για τον οδηγό και για το σύνολο του τομέα και, και επίσης ε, είναι και πιο εφικτό για τις εταιρείε. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον ελάχιστο μισθό και την οδηγία για την απόσπαση. Εμείς πραγματικά θεωρούμε ότι η άλλη πλευρά, αυτοί που καταπολεμούν το κοινωνικό dumping, πρέπει να καταπολεμήσουν την εταιρεία που κάνουν καμποτάζ ε, με το ανατολικοευρωπαίους οδηγούς. Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε. 0% καμποτάζ στη δική μας επιχείρηση. Γι' αυτό λοιπόν ως παρενέργεια αυτού του κανονισμού ο κανονισμός θα σκοτώσει τις διεθνείς μεταφορές. Γι' αυτό αυτή η ρύθμιση των 10 ημερών ε, δίνει επαρκή, περιθώριο στις εταιρείες να βρουν αποτελεσματικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Νίλσεν. Άλλη μια ερώτηση είναι απευθύνω προς το κύριο Ρίπερ. Σκύπερ. Τι πλέον εκτήματα, πιστεύετε ότι θα υπήρχαν, ε, αν υπήρχε μία επίσημη ε, συνεργασία και για τους ελέγχους ε, και για την αλλαγή δεδομένων. Τι πλεονεκτήματα πιστεύετε τα παρουσίαζε μια τέτοια λύση για τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Σκύπερ, Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα, πολλές, πάρα πολλά πλέον εκτήματα η οργάνωση κατάρτισης και εκπαίδευσης, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ε, εντοπισμό περιπτώσεων απάτη στους ταχογράφους, ε, εκπαίδευση για ζητήματα νομοθεσίας, ε, σύνθετης νομοθεσίας. Αυτό ήδη μπορεί να γίνει, αλλά θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν ευρώ ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκή κύκλη μαθημάτων και ε, οργανώσει ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά ε, επιτήρηση. Σας παρακαλώ να κλείνετε σιγά σιγά, λέει η Πρόεδρος. Άρα το σημείο κλειδί είναι η βελτίωση της θέσης ε, πληροφοριών. Θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλά με τις πληροφορίες που έχουμε με τα λίγα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και δεν μπορούμε να μην ελέγχουμε κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Η κυρία Μοντεμοντέρο έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω και τρεις ερωτήσεις προς τον κύριο Πολώνιο. Πρώτα απ' όλα, το τέλος των, των περιορισμών για τα οχήματα χωρίς οδηγό αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νόμου για να εφαρμοστεί αυτή η περίοδος των τεσσάρων μηνών. Τώρα, για την απελευθέρωση του τομέα των μεταφορών. Ε, είναι ήδη απελευθερωμένος ο, ο τομέας αυτός η αγορά αυτή, έτσι. Και υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ό,τι αφορά την πρόσβαση ε, στην, ε, στο επάγγελμα αυτό. Παραδείγματο χάρη, η ενοικίαση, η μίσθωση ε, οχημάτων από εταιρεία που βρίσκεται σε άλλη χώρα για τέσσερι μήνε. Αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλη χρονική περίοδο και μάλιστα είναι κατά των, των ίδιων των εταιριών, κατά των κατασκευαστών, ε, θα αυξηθούν και οι απαιτήσει πρόσβασης. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν αυτοί οι τέσσερις μήνες. Ε, εκτός αν, όπως προτείνεται στην οδηγία για τη μίσθωση χωρίς οδηγό, ακολουθηθεί μια άλλη οδός. Οι διαδοχικές μισθώσεις τώρα, με βάση την υπάρχουσα οδηγία, μπορεί ένα συμβόλαιο ε, να το, το διαδεχθεί ένα άλλο. Ε, τώρα δεν καταλαβαίνω πώς σχετίζεται το άρθρο 5 με την έννοια της σταθερής εγκατάστασης και την πρόταση οδηγίας. Ε, και μια άλλη ερώτηση για την οδηγία σχετικά με την απόσπαση. Ε, αυτό τι επιπτώσεις θα έχει στις περιφερειακές χώρες όπως η Πορτογαλία. Χωρίς μικρόφωνο η απάντηση όμως. Ναι, όπως είπα στην παρουσίαση, η Πορτογαλία έχει μία ε, έντονη δραστηριότητα στις διεθνείς, διεθνείς μεταφορές, όπως και άλλες χώρες, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία. Μιλώντας πάντα, ε, λαμβάνοντας υπόψη είναι το μέγεθος της κάθε χώρας, έτσι. Και αυτό επηρεάζεται, πλήττεται. Ε, ο κατώτατος μισθός του Βελγίου ή της Γαλλίας, της Γερμανίας είναι πολύ υψηλότερος ε, από τον κατώτατο μισθό στις άλλες χώρες που ανέφερα προηγουμένως. Ακόμα και χωρών όπως η Ισπανία. Και αυτό θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλη αύξηση του κόστου. Το διεθνέ εμπόριο ε, αντιπροσωπεύει 35, 30% μάλλον του, του κόστου. Με αύξηση τάξη του 10-15% ε, των μισθών σημαίνει αύξηση 5-10% του συνόλου του κόστου. Ε, και όσοι έχουν τα πράγματα ενώ λείπουν οδηγοί σε όλη την Ευρώπη, το γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις, οι περιφερειακές, θα περιορίζουν τους τόλους τους και περιορίζουν τις μεταφοράς τους σε, σε, μικρές αποστάσεις, ε, αυτό θα οδηγήσει σε πρόβλημα σε ό,τι αφορά ε, το να βρεθούν ε, φορτηγά και βεβαίω μειώνεται, γενικότερα οι μεταφορέ. Παρακαλώ, επόμενο ομιλητή. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και να κάνω μία ερώτηση ε, προ τον καθηγητή από το Κτάντ. Θα ήταν καλύτερο να ε, πάμε να επανέλθουμε στην αρχική έννοια του καμποτάζ, την πρόληψη δηλαδή άδειων ε, φορτηγών που επιστρέφουν στα, σπι... στα... στις πατρίδες τους. Καμία εσωτερική μεταφορά και καμία απόσπαση. Well, uh, Θυμάστε ότι αν είστε μια περιφερειακή χώρα και πρέπει να καλύψετε μια πολύ μεγάλη απόσταση, είναι πολύ δύσκολο για σας να επιστρέψετε εγκαίρως, όπως προτείνεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική αν έχετε μια επιχείρηση σε μια κεντρική χώρα, σε μια χώρα πυρήνα. Επομένως, είναι, δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων. Οι κανόνες αυτοί αναγκαστικά θα εφαρμοστούν διαφορετικά. Και προς τον ε, συναδέλφο από την ε, Σουηδία και προς τον κύριο Παρίλιο να ρωτήσω τι πιστεύουν για τον κύριο Βάμπερερ που ζητά πιο πολύ ευελιξία. Ίσως θα ήθελα να μας απαντήσει ο κύριος από τη Σουηδία πρώτος. Κοιτάξτε, πρέπει εδώ πέρα να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Το είπα και πριν από λίγο, αλλά η ευελιξία αυτή είναι ήδη πάρα πολύ ψηλή σήμερα. δούμε πώς έχει κατάσταση στη Δανία. Όπου έχουμε υπηρεσίες καμποτάζ, καμποτάζ προς την Σουηδία, Σαφώς υπάρχει πολύ ψηλό βαθμός ευελιξίας. Αν δούμε όμως τι γίνεται με τους οδηγούς και τα οχήματα από την Πολωνία, αν δούμε αυτοί σε τι είδους δραστηριότητες, ε, τι είδους δραστηριότητες κάνουν, κάνουν προφανώς καμποτάζ και αυτοί προς τη Σουηδία και προς τη Δανία. Εννοούσα τους χώρους, το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης. Χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης. Εκεί πιο πολύ ευελιξία. Euh, Κοιτάξτε, ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι ο μόνος κλάδος και αυτό απορρέει από μια μελέτη που ζήτησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας κλάδος ο οποίος παρουσιάζει τεράστια ευελιξία, ο πιο ευέλικτος θα έλεγα από όλους τους άλλους τομείς. Και μάλιστα στην ίδια την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήρθε σε εμά τους κοινωνικούς εταίρους, μας είπαν ότι ζήτησαν να γίνει μία μελέτη η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο μόνος κλάδος που ξεπερνά το 48ωρο σε βάση είναι ο τομέας των εμπορευματικών μεταφορών. Μας κάνει εντύπωση που μας ζητάνε αυτή τη στιγμή περισσότερη ευελιξία, μα είμαστε ήδη πάρα πολύ ευέλικτοι. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε και να επιβάλλουμε κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες. Ο κλάδος είναι ήδη πάρα πολύ ευέλικτος, δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερη ευελιξία, αφού είναι αδύνατον. Και να ολοκληρώσω λέγοντα το ακόλουθο. Η Γερμανία, για παράδειγμα, μας λέει ότι τις λείπουν 15 με 30 χιλιάδες χώρες στάθμευσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό dumping δημιουργώντας αυτές τις επιπλέον θέσεις στάθμευσης. Είναι σαν να λέμε ότι για να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες φυλακές. αυτό είναι παράλογο. Ο κύριος Έρντουκ έχει τώρα το λόγο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και να ξεκινήσω με τον κύριο Λάικο. Κύριε Λάικο, για το ερώτημα του ποσοστού καμποτάζ ε, κάνετε. Μας είπατε 0,0% αλλά εδώ πέρα έχω ε, ένα διάγραμμα, ένα χάρτη ε, από την ιστοσελίδα σας ε, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά σε 1.200 τα φορτηγά στη Γερμανία, στην, στον Βασίλειο, 500 στις χώρες Πεντελούξ. Αυτό πώς το δικαιολογείτε λοιπόν αυτές οι πληροφορίες ε, στην ιστοσελίδα μας είναι αληθείς, αλλά 100% των ποσοστών αυτών είναι για διεθνείς ε, μεταφορές, δηλαδή τουλάχιστον να περνάμε ένα σύνορο. Καποτάζ για μένα σημαίνει να κάνει κανείς γερμανικές μεταφορές με φόρτωση και εκφόρτωση στη Γερμανία. Αυτό είναι καποτάζ, το ποσοστό αυτό είναι μηδενικό στην επιχείρησή μας. Άλλη μια ερώτηση προς τον κύριο Σχίπερ. Λέτε ότι το πρόβλημα είναι η εφαρμογή. Εδώ συμφωνούμε. Και αν λοιπόν υπήρξε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ή αν, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν πιο πολλές αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα θέλετε να υπάρξει διεύρυνση των αρμοδιοτήτων από δική σας πλευράς στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είμαι εδώ για να αποφανθώ για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν οι ευρωπαϊκές ε, υπηρεσίες και το τι θα πρέπει να ελέγχεται. Ούτε μπορώ να επισέλθω σε πολιτικά ερωτήματα και θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός γιατί εκπροσωπώ 15 χώρες. Όχι, το θέμα δεν είναι η πολιτική, λέει ο κύριος Έρτογκ. Το θέμα είναι κατά πόσον θέλετε να υπάρχουν πιο πολλές αρμοδιότητες που θα δώσουν δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο αποτελεσματική στην εφαρμογή. Δεν είναι πολιτική ερώτηση. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάντα κάτι το ευπρόσδεκτο, αν έχουμε πιο πολλές δυνατότητες εφαρμογής και ελέγχου. Το θέμα δεν είναι η νομοθεσία όμως, αλλά το πώς συνεργαζόμαστε. Θα πρέπει η, ο έλεγχος και η εφαρμογή να μπει επιτέλους στον 21ο αιώνα. Θα πρέπει να έχουμε πιο πολλές και πιο καλές πληροφορίες, να ανταλλάσσουμε πιο πολλές πληροφορίες και να συνεργαζόμαστε πιο πολύ είμαι με τους ΔΕ για την καταπολέμηση κάποιων μόρφων απάτης και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τσίλε για τρία λεπτά. Ναι, αντί για πινκ πονγκ εγώ προτιμάω το ε, smart tennis. Ε, εν περιπτώσει, εγώ είμαι υπέρ μιας εσωτερικής, μια ελεύθερης αγοράς, ασθενεία αγοράς σε όλους τους τομείς γιατί αυτό μα επιτρέπει να έχουμε ανταγωνισμό με τα διάφορα, μεταξύ των διαφορών κρατών μελών, μεταξύ των διαφορών επιπέδων τη κοινωνία μα κτλ. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο ερώτημά μου αφορά την κυρία Μπερτελό. Αναφερθήκατε στι κοινωνικέ πληρωμέ για άλλε χώρε, για άλλα κράτη-μέλη, εταιρείε που δεν πληρώνουν τι ίδιε εισφορέ, ε, για τις, τις δεξιωτικές φορές, ε, ασφάλιση κτλ. Κοινωνική ασφάλιση. Ε, σας ενδιαφέρουν πιο πολύ οι Λετονοί και οι Πολωνοί συνταξιούχοι ε, ή σας ενδιαφέρουν πιο πολύ, πιο πολύ οι, οι δαπάνες ε, των εταιριών που πληρώνουν ε, τους, ε, και πώς θα πληρώνουν τους οδηγούς τους. Ναι, το σχόλιο που έκανα δεν έχει να κάνει με το επίπεδο των συνεισφορών των εισφορών, αλλά την, την βάση των εισφορών. Διότι εμείς ασχολούμαστε και με το θέμα της αμοιβή. Η αμοιβή δεν είναι μόνο ο μισθός. Είναι αυτό που οι κοινωνικοί εταίροι ονομάζουν ε, το μισθό το διαφοροποιημένο, δηλαδή τη σύνταξη. Βεβαίως πρέπει να επιδείξουμε εδώ καινοτομία. Όταν είμαστε στον ίδιο όμως, ε, στην ίδια αγορά, εντάξει, είναι φιλόδοξο να ζητήσουμε ε, ίδιο μισθό. Διότι υπάρχουν διαφορέ από χώρα σε χώρα, αλλά τουλάχιστον να είναι οι οι επιβαρύνσεις. Να, είναι, να υπάρχει μια ίδια λογική, μια ίδια λογική ένα ίδιο ε, δίκαιο. Ελπίζω να ήμουν σαφή στην απάντησή μου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάποιες χώρες ε, οι βοηθοί ε, λαμβάνουν 10 ε, φορές λιγότερα περισσότερα από άλλους. Ε, είναι πολύ μεγάλες διαφορές, τεράστιες. Εν πάση για τον κύριο Παρίγιο, ε, ποιο είναι το σπίτι του οδηγού, πού πρέπει να πάει μετά από τρεις εβδομάδες δουλειά, ποιο είναι, πού είναι το σπίτι του. Πολύ καλό ερώτημα. Δεν έχουμε απάντηση σε αυτό έως τώρα. Παραδείγματο χάρη, όταν έχουμε έναν οδηγό, Πολωνό, που προσλαμβάνεται από μια πορτογαλική εταιρεία. Πού πρέπει να επιστρέψει. Στην έδρα της εταιρείας στην Πορτογαλία. Αυτό ζητούν κάποιες ομοσπονδίες. Ενώ ο τόπος ε, διαμονής του είναι στην Πολωνία. Η οικογένεια του είναι εκεί. Πρέπει να ζητήσουμε κάποιος να επιστρέψει στην Πορτογαλία να ξεκουραστεί. Στην έδρα που βρίσκεται μια εταιρεία σε ένα, που βρίσκεται σε κάποιο δρόμο, ε, σε κάποιο μεγάλο δρόμο που δεν μπορεί να πάρει καν ποδήλατο. Ε, και εμένα μου αρέσουν πολύ βέβαια, μου αρέσει πολύ η Λισαβόνα με τα δρομάκια τη, αλλά το να έχουμε εταιρείε ε, σε μικρά δρομάκια όπου δεν περνάει καν ποδήλατο, αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για μένα. Λοιπόν, πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα πού βρίσκεται η έδρα, διότι δεν απαντάει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ναι, να πω κάτι. Δεν ξέρω καμία άλλη ευρωπαϊκή νομοθεσία όπου ο πολίτης πρέπει να πάει σε ένα συγκεκριμένο μέρος μετά από τρεις εβδομάδες. Ε, ε, υποχρεωτικά. Μάλιστα, να συνεχιστεί η συζήτηση. Ο κ. Πάβελ Τερλίντσκα έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι βλέπω πολύ προστατευσμό στην Ευρώπη αλλά και πολλές αθέμενε πρακτικές ε, κύριε Μπερτελό, μπορείτε να μου πείτε το μέσο μισθό και το πώς διαρθρώνεται για έναν καλό οδηγό. Αυτό αναφέρεται στο τελευταίο γράφημα που δημοσίευσα. Όλα μαζί, μαζί με τις εισφορές δηλαδή, το, το μέσο κόστος της ώρας οδήγησης είναι 30 ευρώ περίπου ο μέσος οδηγός έχει ένα μέσο μισθό καθαρό 2.200 ευρώ. Ε, ευχαριστώ. Δεν είναι σωστή αυτή η πληροφορία. Αυτός είναι ο μέσος όρος ενός τσέχου οδηγού και από ό,τι κατάλαβα τα στοιχεία είναι πολύ συγκρίσιμα. Ε, δεύτερον, είπατε μια σειρά από πράγματα, αλλά ποιος είναι ο σκοπός, ποιος πρέπει να είναι ο σκοπός που πρέπει να επιτευχθεί με το πακέτο κινητικότητας. Ευχαριστώ που θέλετε το ερώτημα αυτό. Σε ό,τι αφορά το καμποτάζ, εμείς είμαστε κατά. Κατά οποιασδήποτε απελευθέρωση του καμποτάζ. Το να πάμε στις πέντε μέρες χωρίς όριο ε, ε δραστηριότητας ε, ε, αυτό ουσιαστικά είναι μια μεταφιεσμένη απελευθέρωση ε, χωρίς να υπάρχει μια περίοδος ε, ξεκούραση μεταξύ δύο περιόδων του καμποτάζ. Δεν μπορεί το καμποτάζ να γίνει ουσιαστικά να, να οδηγήσει στην παράκαμψη των κανόνων της ιστορικής αγοράς. Συγγνώμη, χάνετε, χάνετε χρόνο στο ερώτημά μου, είναι σαφές. Ποιος είναι ο στόχος του πακέτου κινητικότητας. Δεν μου απαντήσετε. Οπότε το επόμενο ερώτημά μου, ποια είναι η διαφορά σύμφωνα με το δικό σας, τη δικό σας προοπτική ανάμεσα στις τρεις και τις πέντε μέρες και πώς το όριο των τριών μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς, τις μεταφορές. Ακούστε, ο στόχος δεν είναι να παρεμποδίσουμε τις διεθνείς μεταφορές. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε το, το να περνάμε τα σύνορα να οδηγήσει σε ο στόχο μάλλον του πακέτου, για να είμαι πολύ συγκεκριμένο, να απαντήσω στο ερώτημά σα κύριε, είναι να μην έχουμε ένα αυτόνομη αγορά που να μην συνδέεται με καμιά εμπορική ε, σχέση. Διότι εδώ έχουμε μια εμπορική σχέση μεταξύ ενό πελάτη και του πελάτη αυτού του πελάτη ε, και δεν είναι μια αυτόνομη αγορά που κάποιοι βρίσκονται σε μια χώρα μόνο και μόνο ε, για να πάρουν αγορές χωρίς να έχουν συμβασιακή ε, σχέση. Δεν έλαβα απάντηση. Εγώ ρώτησα τη διαφορά μεταξύ των τριών και των πέντε ημερών. Ε, εσείς μου είπατε τι είναι το καμποτάς, τι δεν είναι. Εγώ δεν είμαι υπέρ των αθέμητων πρακτικών. Αλλά έθεσε ένα ερώτημα και δεν έλαβα απάντηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τελίτσκα ήταν λοιπόν που μίλησε και τώρα είναι η σειρά μου. Λοιπόν, Θέλω να ρωτήσω πρώτα τον καθηγητή, τον κύριο Μπροκόφσκι. Μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε αυτό που είπατε. Είπατε ότι χοντρικά χρειάζονται κανόνες διαφορετικοί μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Είπατε αυτό. Απαντάτε με ναι ή με όχι. Αυτό λέτε. Είναι έτσι. Κατάλαβα καλά. Όχι. Εγώ μόνο είπα ότι επηρεάζονται διαφορετικά οι νέοι κανόνες, οι χώρες της ε, Κεντροανατολικής Ευρώπης σε σχέση με τις χώρες του πυρήνα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θέλετε να υπάρξει μια διόρθωση έτσι όλοι να υπάρχει εξίσωση προς τα πάνω. Δηλαδή οι κοινωνικοί κανόνες ε, να εξισωθούν προς τα πάνω. Συμφωνείτε φαντάζομαι. συμφωνείτε να υπάρχει ίση αμοιβή για ίση εργασία. Διότι αυτό δεν το άκουσα να το λέτε. Εσείς θεωρείτε ότι εάν βάλουμε ίσο μισθό για την ίση εργασία ε, πάμε προς μια ίση ε, μεταχείριση των εργαζομένων στην Ευρώπη. Αν όλα τα άλλα είναι ίσα, όπως το κόστος ζωής, ναι. Ένα άλλο ερώτημα τώρα. Αλλά μιλάει πρόεδρος, έτσι. Κύριε Παρίγιο, είπατε το θέμα του ελέγχου και της απάτης είναι κρίσιμο σε αυτό το πακέτο. Θα ήσασταν υπέρ να υπάρχει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ή μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων να εξασφαλίσουμε επιτέλους ότι θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ναι, βεβαίως, τρεις φορές ναι. Με ένα στοιχείο μόνο, διότι είναι εδώ και το ECR, όταν λαμβάνουν έλεγχοι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τα 100 οχήματα, τα 30 παραβιάζουν τον νόμο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα στην Ευρώπη, στα 2.400.000 φορτηγά που κυκλοφορούν κάθε μέρα, υπάρχουν 700.000 οχήματα τα οποία ε, είναι παράνομα. Εάν δεν έχει καταλάβει η Κομισιόν ότι πρέπει να πάρθουν αυστηρά μέτρα, νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Μάλιστα, ευχαριστώ τον κύριο Παρίγιο. Και επαφήνομαι στο ECR. Ε, είστε και εσεί υπέρ μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για, τα οδικ... για οδικές μεταφορές που να ελέγχει πραγματικά. Νομίζω ότι η ερώτηση αυτή είναι μια ερώτηση δύσκολη για μένα. Δεν μπορείτε να απαντήσω. Είναι πολιτική. Νομίζω ότι και η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί επίσης να λειτουργήσει καλά. Και τελευταίο ερώτημα. Θα τη θέσω και στον κύριο Παρίγιο. Με κόψατε. Αν προσθέτω 14 λεπτά. Κύριε Παρίγιο, θέλω να πείτε, να καταλάβω, δώστε να καταλάβω, ποιο είναι το καθεστώς όλων αυτών των οδηγών που ε, ε, προσλαμβάνονται σε εταιρείες ταχυδρομικές θηρίδες και δεν ε, εργάζονται στις χώρες τους. Ε, ποιο είναι το καθεστώς τους. Να σας πω. Είναι μοντέρνοι σκλάβοι σε μια μοντέρνα Ευρώπη. Και λέει, προσέχω τις λέξεις μου, έτσι, όταν έχουμε οδηγούς Ρουμάνους που εργάζονται μήνες και μήνες στο Βέλγιο και στη Γαλλία με ένα καθεστώς σλοβάκικο, μόνο σκλάβου μπορώ να του ονομάσω. Δεν είναι αποσπασμένοι. Το άρθρο 1 τη οδηγία για την απόσπαση αναφέρει ότι δεν μπορεί κάποιο να αποσπαστεί από την συνηθισμένη χώρα εργασία του. Ο κύριος Πίτερ Λούγκριν τώρα έχει το λόγο. 3,5 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βλέπουμε λοιπόν για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί, γιατί ουσιαστικά απαρτίζεται από πολλούς διαφορετικούς κανόνες των διαφορετικών κρατών μελών. Δεν έχουμε το ίδιο κοινωνικό επίπεδο, δεν έχουμε το ίδιο οικονομικό επίπεδο, αν ήταν όλα ευθυγραμμισμένα, μπορεί να λειτουργούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρει να λειτουργήσει αποτελεσματικά ούτε στο μέλλον. Ας δούμε τι γίνεται για παράδειγμα στη Σουηδία, στον Καποτάζα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι στην Σουηδία αυτή υπάρχουν χιλιάδες φορτηγά από το εξωτερικό που κάνουν καμποτάζ σε αυτή τη χώρα. Προέρχονται από άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδίδονται σε καμποτάζ στην επικράτεια της Σουηδίας. Και αυτό γίνεται βέβαια με την ίδια την τη βοήθεια και την υποστήριξη της οδηγίας για το καμποτάζ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ απασχολήθηκα στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές για πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν. Όταν λοιπόν ακούω συναδέλφους να λένε ότι δεν ασχολούνται με το καποτάζ, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχω ακούσει ποτέ. Για παράδειγμα, εσείς μας λέτε ότι έχετε ένα γραφείο, μη στη Γερμανία, έτσι δεν είναι. Επομένως, τα γερμανικά φορτηγά με γερμανικές πινακίδες στους Γερμανούς αυτούς οδηγούς δίδεται πραγματικά ένα μισθό γερμανικό ή όταν απασχολείται οδηγούς από άλλες χώρες διατηρείται την αμοιβή αυτή της Γερμανίας. Σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Ναι, κοιτάξτε λίγο και την ιστοσελίδα μας. Έχουμε μια θηγατρική στη Γερμανία, αλλά αυτό ουσιαστικά απασχολεί μόνο κάποιες ομάδες εργαζομένων που ασχολούνται με τις πωλήσει. Και είναι Γερμανοί εργαζόμενοι αυτοί, δεν κάνουμε καμποτά στη Γερμανία. Η ομάδα πωλήσεων απλώς βρίσκεται σε αυτή τη θηγατρική και κανείς άλλος. Αν λοιπόν εντοπίσετε κάποιον δικό μα να κάνει καμποτάζ σε άλλη χώρα, στη δική σα τη χώρα για παράδειγμα, στείλτε μου μια φωτογραφία και θα το διευθετήσω. Εγώ είμαι επικεφαλή αυτή τη επιχείρηση, ξέρω πολύ καλά γιατί μιλάω. Ναι, ναι, ωραία. Και αυτή η επιχείρησή σα, λοιπόν υποβοηθείται από μία άλλη επιχείρηση επενδυτική, έτσι δεν είναι, και νομίζω ότι εσείς καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αυξήσετε το κόστος σας. Τα φορτηγά λοιπόν αυτά, τα οποία έχουν γερμανικές πινακίδες και που έχουν ε, Γερμανούς οδηγούς δεν τα χρησιμοποιείτε πουθενά ούτε στις κάτω χώρες. Νομίζω ότι πηγαίνετε στις κάτω χώρες και εκεί πέρα δίδετε μισθό κάτω χωρών, έτσι δεν είναι νομίζω ότι στέλνετε βασικά τα φορτηγά σας παντού στην Ευρώπη και δημιουργείτε έναν αθέμητο εσωτερικό ανταγωνισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζετε τα πράγματα πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι, αλλά στην πραγματικότητα αυτό κάνετε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω καθόλου τι με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, γιατί ο ορισμός του καποτάζ είναι σαφής. Ξένος οδηγός με ξένο φορτηγό που κάνει εγχώρια μετακίνηση, εγχώρια μεταφορά αυτό δεν μας αφορά μας καθόλου. Ξέρετε ότι εμείς ε, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι καμποτάζ του να φέρεστε βασικά σε διεθνείς μεταφορές. Μεταφορές από την Ουγγαρία στη Γερμανία με γερμανικά φορτηγά. Η κυρία Αγνουτού έχει το λόγο. Το πρώτο ερώτημα προς τον κύριο Σίπερ μα είπατε ότι έχουμε ένα ποσοστό 20 με 30% αφορά την απάτη, απάτη ταχογράφου. Δεν πιστεύετε ότι ε, εφόσον ε, αποδειχθεί λοιπόν η απάτη αυτή και εφόσον ε, ο οδηγός δεν έχει τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει τουλάχιστον να κινητοποιηθεί το όχημά του ή να επιβληθούν σημαντικές χρηματικές ποινές προκειμένου να πείσουμε τελικά την επιχείρηση μεταφορά να συμμορφωθεί. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. <clears throat> Er ναι, θα πρέπει να υπάρχουν ε, κυρώσεις και υπάρχουν αιτήματα για κυρώσεις ε, σωστές και αναλογικές, ε, οι οποίες θα αποτελούν αντικίνητρο. Αλλά σε ό,τι βλέπουμε, σε ό,τι παρατηρούμε, είναι ότι με την απάτη βγαίνουν πολλά χρήματα. Με ένα φορτηγό μπορούμε να βγάλουμε 10.000 ευρώ παραπάνω κάθε χρόνο. Και έτσι λοιπόν ε, ο επιχειρηματίας που τα βάζει κάτω λέει κοιτάξτε να δείτε αξίζει τον κόπο, θα το κάνω. Θα κάνω την απάτη και θα πληρώσω και το πρόστιμο όποτε μου έρθει. Το σύστημα λοιπόν ε, βασίζεται και στην καλή φήμη η οποία θα μπορούσε να αποτελεί επαρκές κίνητρο για να καταργηθεί για παράδειγμα η άδεια ενός ε, επιχειρηματία. Ευχαριστώ. Το δεύτερο ερώτημά μου αφορά την κυρία Μπερτελό. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Θα ήθελα να έχω και την παρουσίασή σας αν γίνεται. Προηγουμένως είπατε πολύ σωστά, δηλαδή δεν μίλησατε για προστατευτισμό ακριβώς, αλλά εγώ νομίζω ότι με έναν έξινο προστατευτισμό μπορούμε να βρούμε λύσεις. Βεβαίως το κόστος ζωής δεν είναι το ίδιο από μια χώρα στην άλλη. Αλλά αν χρησιμοποιούμε συνέχεια αυτό το επιχείρημα, δεν πρόκειται ποτέ να επιληθεί αυτό το ζήτημα θέμη του ανταγωνισμού. Εγώ πιστεύω ότι αντιθέτω χρειάζεται ένα έξυπνο προστατευτισμό. Για να αποφύγουμε λοιπόν την εκμετάλλευση τη μισθολογική που επιτρέπει η παρούσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν πιστεύετε ότι η απλή αρχή ίση εργασία ε, για ίσο μισθό, ίσο μισθό για ίση εργασία, να εφαρμόζεται για όλα τα κράτη-μέλη. Παρότι συμφωνώ με τον συνάδελφο Λούνγκριν, ότι η σημερινή συζήτηση δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί καλά ε, και σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Ακούστε, εμεί διαπιστώνουμε ότι υπήρχε μια ανάγκη. Τα κράτη-μέλη, πριν ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βάλει μια πρόταση, έχουν ατομικά προβλέψει εθνικού κανόνε. Η Γερμανία πρώτα, μετά η Γαλλία και άλλε η δυσκολία για την εφαρμογή της απόσπασης. Και σας, εγώ σας το λέω αυτή αρχής, η απόσπαση για μας δεν είναι κάποια καταπληκτική ιδεώδης λύση. Είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στον τομέα των μεταφορών. Αλλά δεν έχουμε κάτι άλλο, αυτό έχουμε. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για την κοινωνική κατάσταση των οδηγών. Προσοχή λοιπόν, προσοχή. Όταν λέμε ίση εργασία, ίση αμοιβή, μετά όμως λέμε ίσο, ίσο έδαφος, ίσο μισθό. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε σε εδάφη εδώ. Είμαστε σε ροές. Υπάρχει μια ροή. Ευχαριστώ την κυρία Μπερτελό. Ο κύριος Ντέλη έχει το λόγο για δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο σύντομες ερωτήσεις προς την κυρία Μπερτελό. Διάβασα στις εφημερίδες χθες ότι εκατοντάδες φορ... Ναι, φορτηγατές έκλεισαν τα σύνορα με την Ιταλία και το Βέλγιο δεν ήταν, δεν ήταν ικανοποιημένοι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πώς θα τους προστατεύσει από τις ανατολικές χώρες με τον, στον ανταγωνισμό τους με το χαμηλό κόστος. Εντάξει, βεβαίως ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί, αλλά πιστεύετε ότι να μπλοκάρει κανείς τους δρόμους είναι ένα σωστός τρόπος για να προστατεύσουμε την στενή ιστορική αγορά μεταφορών. Ε, λίγο προκλητικά έτσι το θέλω το ερώτημα. Τώρα ένα δεύτερο πιο σοβαρό. Αναφερθήκατε στη διαφορά μεταξύ μισθών ε, από χώρα σε χώρα. Ε, ειλικρινά πιστεύετε ε, ότι αυτές οι διαφορές θα απαλληφθούν εφόσον ε, ακολουθούν οι κανόνες για την απόσπαση των εργαζομένων και τι γίνεται με τις άλλες, ε, άλλους τρόπους μεταφοράς, τα αεροπλάνα και τα τρένα, διότι και εκεί έχουμε διεθνές, διεθνείς μεταφορές και εκεί υπάρχει το θέμα της ίσης αμοιβή για ίση εργασία. Ε, αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ για το ερώτημα, για το πρώτο. Ε, σας σας ε, παραπέμπω μάλλον στον, τον, στον διπλανό μου. Η ETF είναι αυτή που μπλόκαρε ε, δεν καταλαβαίνουμε βέβαια ήδη το, όλοι το ίδιο για το τι συνέβη στις 23 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων. Νομίζω ότι υπάρχει μια ε, παρανόηση. Εφαρμόζεται η απόσπαση στο μέρο μεταφορών παρότι αναμένοντας ε, μια ήδη λέξη σπεσιάλης θα εξακολουθεί να ισχύει ε, η νομοθεσία του 93 τώρα για τους μισθούς. Ε, το να του βάλουμε να έχουν όλοι το ίδιο μισθό και ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα αγωνισμού στην Ευρώπη, εντάξει, δεν είναι ουτοπία. Τι διαπιστώνουμε όμω, Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν εταιρείε που έχουν ένα πλεονέκτημα ανταγωνιστικό, διότι υπάρχει διαφορά και στους μισθούς και στις εισφορές. Είναι στην ίδια, θέση ανταγωνισμού? Όχι. Δεν υπάρχει όμω κάποια ιδανική λύση. Εμεί έχουμε μια φιλόδοξη, ένα φιλόδοξο καθεστώ για αυτό, το, για να δημιουργήσουμε ένα καθεστώ για τον κινούμενο, μετακινούμενο εργαζόμενο, λέμε είμαστε μακριά από αυτό. Του επόμενου μήνε λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το εναρμονισμένο αυτό καθεστώ, το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε για τον διεθνή οδηγό. Είναι μια δύσκολη συζήτηση και ψάχνουμε λύσει όλοι μαζί από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, δυστυχώ είναι ο χρόνο. Ιζαμπέλα Ντεμόντε, δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Παρίλο. Σε σχέση με τον χρόνο οδήγηση και ανάπαυση, η υφιστάμενη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μια άλλη διάρθρωση των εβδομάδων και προβλέπει στη συνέχεια συγκεκριμένου χρόνους ανάπαυση. Ποια είναι η άποψή σα, ανταποκρίνεται πραγματικά αυτό στι ανάγκε οδική ασφάλεια, βοηθά στο να υπάρχει καλύτερη εξορρόπηση προσωπική και επαγγελματική ζωή διασφαλίζεται η καλύτερη ανάπαυση των οδηγών και τι προβλήματα βλέπετε εσεί να αναδύονται από την πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Για τον πολύ απλό λόγο ότι όταν τροποποιούμε τον χρόνο οδήγηση και τον χρόνο ανάπαυση, όπως είπα και στην παρέμβασή μου, τότε όλοι οι κανόνες και όλα τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία εξαρτώνται από αυτό τροποποιούνται και αυτά με τη σειρά τους. Τροποποιώντας λοιπόν το χρόνο ανάπαυσης και οδήγησης, τροποποιούμε το χρόνο εργασίας. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και προσέξτε πραγματικά τι λέω, έκανε μία πρόταση λέγοντας ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Και αυτό που ακούμε σήμερα είναι ότι πρέπει εκ νέου να τροποποιήσουμε το σύνολο του χρόνου οδήγηση, αν είναι να συμμορφωθούμε τελικά με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί είμαστε κατά αυτού. Θεωρούμε ότι το υφιστάμενο καθεστώ θα πρέπει να παραμείνει ω έχει. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι οι υφιστάμενοι κανόνε να εφαρμόζονται. Όχι να τροποποιούμε του κανόνε που δεν καταφέρουμε να του επιβάλλουμε. Μάλιστα. Σε σχέση με το ζήτημα της ευελιξίας και την επιστροφή στην κατοικία. Ως προς αυτό υπάρχει τώρα μία συμφωνία, έτσι δεν είναι. Και προβλέπεται επίσης και η δυνατότητα ανάπαυσης στο θάλαμο οδήγησης. Συμφωνείτε εσείς να πούμε ότι όλες οι διεθνείς μεταφορές και οι μεταφορές καμποτάζ θα πρέπει να υπάγονται στο καθεστώς καταγραφής μεσοταχογράφου. Εμείς είμαστε κατά της ανάπαυσης μέσα στο όχημα. Δεν μπορεί να καταμετράται έτσι η εβδομηδία περίοδος ανάπαυσης. Επίσης, Ετίθετο επίσης και ο κανονισμός και η εφαρμογή του κανονισμού του 2006 που λέγεται ότι κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης ο οδηγός είναι ελεύθερος να κάνει όποια μετακίνηση θέλει. Δηλαδή δεν έχει σαφώ την υποχρέωση να μείνει μέσα στο όχημα κατά τη διάρκεια τη ανάπαυση. Τώρα υποχρεώνουμε τον οδηγό να παραμείνει μέσα στο όχημα. Για μας λοιπόν είναι αδύνατον ο οδηγός να μένει μέσα στο όχημά του προκειμένου να παυθεί για τις 45 ώρες που προβλέπονται. Επόμενος ο μελητής παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχόλια προς τον κύριο Φασκόφσκι, επιτρέψτε μου. οι υπηρεσίε μεταφορών θα είναι πιο ακριβέ, αλλά παντού ίδιε. Ε, κάπου λιγότερο, κάπου περισσότερο. Σε ποιο κράτος μέλος θα υπάρχουν ε, πιο πολλέ μικρομεσαίες επιχειρήσει από τι καινούργιε, φυσικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, φυσικά. Θα είναι πιο ακριβές ε, στα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία εξαρτώνται πιο πολύ από τις μεταφορές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη προφανώς. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις μεταφορών θα χαθούν από την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Σλοβακία, όπως και στη Βουλγαρία. Σας ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς την κύριο Πολωνία, τώρα. Πόσες ημέρες χρειάζεται ένα οδηγό ε, για να πάει από την Πορτογαλία, από τη μέση τη Πορτογαλία μέχρι τη μέση τη Γερμανία. Πόσε μέρε χρειάζεται? Eh, Έχουμε περίπου 9.000 φορτηγά τα οποία διανύουν τα σύνορα μας κάθε μέρα. Η Γερμανία προφανώς ε, αποτελεί το 1 τέταρτο, το 1 πέμπτο της αγοράς ε, προορισμού μας, αν θέλετε. Άρα είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμα. Πολλοί από αυτούς που εκφορτώνουν στη Γερμανία έρχονται στην Πορτοκαλία για να φορτώσουν στην Ισπανία ή, σε κάποιο, ή στην ε, Πορτογαλία, στην Ιβρική Χερσόνησο. Είναι κλασική αυτή η σε καποιο στην πορτοκαλια στην ιβρικη χερσονησο ειναι κλασικη αυτη η συμπεριφορα για τις φορτώσεις, εκφορτώσεις στην Γερμανία και στην Πορτοκαλία Το θέμα είναι το πόσο παίρνει, πόσες μέρες παίρνει αυτό το ταξίδι. Ναι, αυτό θα έλεγα αυτό θα ήθελα να πω. 45 ώρες. Δύο σύντομες περιόδοι ανάπαυσης και αυτό είναι κακό για τον οδηγό. αν φύγει κανείς από την Ισπανία, πάει στη Γερμανία, εκφορτώσει και μετά ξαναπάει στην Ισπανία σε κάποιες περιπτώσεις ε, μπορεί να πάρει 45 ημέρες η, η επιστροφή στη χώρα του καθενός. Ο κανόνας λοιπόν αυτό θα πρέπει να τραπαποιηθεί και θα πρέπει να καταστεί δυνατόν σε μία περίοδο τέσσερα εβδομάδων να έχει κανείς δύο-τρεις πιο σύντομες περίοδους αναπαύσης, η οποία θα αποζημιώνεται με μία πιο μακρά εβδομηδιαία ανάπαυση κοντά στην κατοικία του καθενός. και έχουμε διάφορους υπαλληλούς ε, μετανάστες στην Πορτογαλία. Και θέλουν προφανώς ο χώρος αναπαύσης να είναι στην οικογένειά τους. Ευχαριστώ. Δεν είχα φανταστεί ότι θα απαντούσατε τόσο πολύ ώρα σε ένα τόσο απλό ερώτημα και δεν έχω πλέον χρόνο για να σχολιάσω. Λυπάμαι τρία μισή λεπτά ο καθένας. Ε, ξέρω είναι λίγο έτσι ενοχλητικό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Κυρία Μάισνερ, θα δώσετε το λόγο στον κύριο Τελίτσκα. Τι καλή που είστε. Κύριε Τελίτσκα, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ναι, ακούστε, θα χρησιμοποιήσω τα ερωτήματα της συναδέλφου της κυρίας Σασκούμπιλμπάου δεν μπορείς να είναι εδώ σήμερα αλλά το ερώτημα όμως είναι, επανέρχεται και είναι το ίδιο ουσιαστικά απλώς αυτή τη φορά θα ζητήσω από την κυρία Μπερτελό ή σε κάποιον άλλον να μου πει εν συντομία τι είναι αυτό που αιτιολογεί ε, σε ποιες περιπτώσεις το καμποτάζ και γιατί. την απαγόρευση του καμποτάζ μάλλον. Ναι, να σας απαντήσω. Η διάρκεια, για τη διάρκεια του καμποτάζ, η διάρκεια του καμποτάζ μπορεί να είναι maximum τρει ημέρε. Πρέπει να μπορεί κάποιο να κάνει μια εσωτερική μεταφορά μετά από μια διεθνή μεταφορά. Έτσι όπω το βλέπουμε εμεί, ε, για να μπορέσει να επιστρέψει κάποιο στη βάση του. Είναι το ίδιο ερώτημα για όλους. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η διαφορά και ποια είναι η διαφορά στην αιτιολόγηση επίσης. Ναι. Er ήθελα να πω ότι ο στόχος ε, είναι να μην χρειαστεί κανείς να επιστρέψει με το φορτηγό άδειων. Αυτό δεν είναι καλό το και το περιβάλλον εκατοντάδες χιλιόμετρα άμα ε, άδειος. Μιλάμε για εθνικές μεταφορές, αλλά τρεις ημέρες ε, αρκούν. Φτάνουν και περισσεύουν. Δεν ξέρω αν μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημα στα αγγλικά, αν γίνεται. Ναι, βεβαίω. Ποια είναι η κατάλληλη διάρκεια για το καμπετέζ, καμποτάζ στο νέο πακέτο και γιατί. Εμείς θεωρούμε ότι το καμποτάζ ρυθμίζεται πολύ σωστά αυτή τη στιγμή. Με, τον με την τεχνική έννοια του όρου, έτσι, στην ίδια χώρα. Επτά μέρες είναι μια καλή διάρκεια. Εμείς δεν συμφωνούμε με την πρόταση αλλαγή. Και κάτι που δεν έχει καταλάβει κανείς νομίζω, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η αλλαγή στην ομοθεσία του καμποτάζ δεν μας αφήνει να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καμποτάζ ε, για τρεις μέρες και να επιστρέψουμε άδειοι. Ε, αυτή η επιχείρηση καμποτάζ συχνά ε, οδηγεί στο να φτάνουν άδεια φορτηγά στη Γαλλία, παραδείγματο, χάρη, από την Αγγλία και πάει από την Βόρεια Γαλλία ε, στον Μπορντό και μετά στην Ισπανία, διότι δεν υπάρχουν πάντα εμπορεύματα για την Ισπανία. Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία αυτό θα απαγορεύεται. Ο κύριος Τέιλορ έχει το λόγο τώρα. Παρακαλώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι ε, σύντομο. Δύο ερωτήσει. Για τον κύριο Παρίγιο. Ποια είναι η αντίδραση της ETF ε, σε ό,τι αφορά ε, τα ξενοδοχεία και το πάρκινγκ από μη οργανώσει οργανώσεις η παροχή αυτών των ε, υπηρεσιών. Θα, θα θέλετε να αναπτύξετε μια τέτοια ιδέα, να την προωθήσετε. Δεύτερον, ε, ποια θα είναι η αντίδραση της CTF στην ιδέα οι εργοδότες να στέλνουν οδηγούς αντικατάστασης για να μπορέσει να συνεχίσει το φορτηγό το δρόμο του και ο οδηγός, ο, ο πρώτος, να επιστρέφει πίσω σπίτι του να ξεκουράζεται. Νομίζω πως είναι μια επικοδομητική λύση. Πώς το βλέπετε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Για το πρώτο, για την επιστροφή στην έδρα, για τον εργοδότη δηλαδή που θα στείλει έναν άλλον οδηγό αντικατάστασης. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, ο οδηγός επιστρέφει στη χώρα του με έξοδα της επιχείρησης. Αυτό που θέλουμε εμείς, μία από προτάσεις που ακούσαμε στο κοινωνικό διάλογο, είναι να επιστρέψει στη χώρα που είναι, βρίσκεται η έδρα της εταιρεία. Αυτό βέβαια είναι παράδεκτο, Είναι εκτροματικό. Σας έδωσα ένα παράδειγμα με την πολλαλική εταιρεία για τον Πολωνό οδηγό. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να νομιμοποιήσουμε αυτό που ισχύει σήμερα. Η επιστροφή στη χώρα διαμονής του οδηγού να γίνεται με έξωτα της επιχείρησης, όπως ισχύει σήμερα. Αλλά αυτό δεν έχει νομιμοποιηθεί. Εμείς θέλουμε να νομιμοποιηθεί αυτό, να κωδικοποιηθεί. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε κάποια άλλη κατεύθυνση όπου θα πρέπει ο οδηγός να αναλάβει ο ίδιος το έξοδο αυτό. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να πράξει. Ναι, αλλά γιατί να επιστρέψει και το φορτηγό. Γιατί να μην επιστρέψει ο οδηγός και να συνεχίσει το φορτηγό. Και να απαντήσετε και στο ερώτημά μου για τις κοινωνικές εταιρείες ε, μη κερδοσκοπικές για το πάρκινγκ και το ξενοδοχείο. Ναι, ακούστε, για μας το όχημα πρέπει η ουσιαστική του, η ουσιαστική του δραστηριότητα ε, να γίνει στη χώρα που είναι καταγεγραμμένη η εταιρεία. Δεν γίνεται να έχουμε μια εταιρεία που εγκαταστάται σε μια χώρα και τα οχήματα να μην εργάζονται, να μην δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε εκείνη τη χώρα. Εκεί αρχίζει το κοινωνικό ντάμπινγκ και αυτό με τους ανταγωνισμούς. Η δραστηριότητα λοιπόν της εταιρεία, ένα ουσιαστικό μέρος αυτής, πρέπει να λαμβάνει χώρα εκεί όπου είναι ε, η έδρα της. Τώρα για το πάρκινγκ. Ε, ακούστε, τα πάρκινγκ δεν υπάρχουν για να κοιμούνται οι οδηγοί. Τα πάρκινγκ υπάρχουν για να σταματήσει ένα όχημα, να μπορέσει να, κάνει, να πληθεί ο οδηγός, να φάει κάτι και να ξαναφύγει. Το πάρκινγκ λοιπόν δεν είναι τόπος όπου μπορεί κάποιο να μείνει, να ζήσει. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Όχι, το ερώτημά μου είναι ξενοδοχείο, ξενοδοχείο και πάρκινγκ. Ξενοδοχείο και πάρκινγκ και για τον οδηγό και για το ε, αυτοκίνητο. Γιατί να μην γίνει αυτό μέσω μιας διευκόλυνσης από μια εταιρεία με καταστροφικό χαρακτήρα. Ναι, κλείστε παρακαλώ. από τη στιγμή που απαγορεύεται να ξεκουραστεί κάπως εβδομαδιαίως σε ένα πάρκινγκ, πρέπει ο εργοδότης να φροντίσει ο οδηγός να ξεκουραστεί σε ένα μέρος ε, ε, που να πληρεί τις προϋποθέσεις, ξενοδοχείο, δεν ξέρω. Είναι φυσιολογικό πάντως ένας οδηγός να μπορεί να ξεκουραστεί σε ένα μέρος λίγο πιο μεγάλο από δύο τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Μπακ τώρα πρέπει να πάρει το λόγο ή ο κύριος Λούγκριν θα αντικαταστήσει τον κύριο Μπαχ, ή τον κύριο Μπαχ μάλλον πρώτος γιατί πρόκειται να αποχωρήσει. Λούγκριν, εσύ θα μείνετε λίγο ακόμα μαζί μας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να σας ακούσουμε τον κύριο Μπαχ τότε πρώτο. Και έχετε δυόμιση λεπτά. Δυόμιση λεπτά και θα είμαι αυστηρή. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είστε πάρα πολύ ευγενικοί και ιδιαίτερα ευέλικτοι μαζί μου και να ευχαριστήσω βέβαια και του συναδέλφου για την ευελιξία του. Δύο ερωτήσει. Η πρώτη απευθύνεται στον κύριο Σκύπερ όσον αφορά τι εικονικέ αυτέ εταιρείε γραμματοκιβωτίου. Τι πιθανότητε πιστεύετε ότι υπάρχουν να ρυθμίσουμε πιο αυστηρά προκειμένου να καταφέρουμε να περιορίσουμε κάθε κατάχρηση που γίνεται μέσω των εικονικών αυτών εταιριών. Δεύτερο ερώτημα για τον κύριο Παρίγιο. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια μεταφατική ε, φάση, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εσείς δεν δέχεστε με τίποτα οποιαδήποτε ανάπαυση στον θάλαμο οδήγηση. Ενδεχομένω αν είχαμε ένα κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένε υποχρεώσει για τα κράτη-μέλη να δημιουργηθούν δηλαδή ασφαλείς χώροι στάθμευσης, να προβλεφθούν όλες οι απαραίτητες άλλες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσατε εσείς να δεχτείτε ενδεχομένως να υπάρξει μία μεταβατική φάση. Σας ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. μιλήσω Ολλανδικά καλύτερα. Θα κοιτάξω το πώ, όχι το τι. Πιο αυστηροί κανόνε, πιο αυστηροί κανόνες. Αν θέλουμε καλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία, αν θέλουμε να υποστηρίξουμε μεν του ΔΕ και να έχουμε πιο πολύ έλεγχο στι εθνικέ ε, αυτέ δραστηριότητε, μπορεί να κάνουμε πολύ πιο πολλά και με την ήδη υφιστάμενη νομοθήση. χρειάζεται απλά καλύτερη συνεργασία στο σημείο αυτό και η πιο αυστηρή νομοθεσία θα μπορούσε να βοηθήσει ενδεχομένω. Κοιτάξτε, εμείς στην ETF παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά αυτά που έχουν να πούνε οι, οι οι καλοί εργοδότες, αν μου το επιτρέπετε, οι οποίοι μας λένε ότι θα μπορούσαν εύκολα, αν υπάρχει ο σωστός σχεδιασμός και τα σωστά μέσα, τότε να μπορούν να επιστρέφουν και να εξεκουράζονται στα σπίτια τους οι οδηγοί. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι είναι θέμα καλύτερης οργάνωσης και όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο, γενικά ξέρετε οι μεταβατικές περίοδοι δεν είναι καλές για κανέναν. Λίγα δευτερόλεπτα έχω ακόμα. Μία ερώτηση προς την κυρία Μπερτελό. Μία επέκταση του καμποτάζα θα ήταν δυνατή. Είδαμε και μία γραφική παράσταση δική σας με κάποια παραδείγματα για την εσωτερική αγορά και τις εθνικές αγορές Προβλέπετε, πιστεύετε ότι μια τέτοια επέκταση θα ήταν ίσως πιο δύσκολη για τις εθνικές αγορές, μια επέκταση του καμποτάζα. Η απάντηση είναι σαφώς ναι. Γιατί ακόμα και με την πλαισίωση που ξεκίνησε το 2009 δεν καταφέραμε να περιορίσουμε την αύξηση του καμποτάζ και τις επιπτώσεις του στις εθνικές εσωτερικές αγορές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ας περάσουμε τώρα στην φυσιολογική ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Λούγκριν, αντικαθιστάτε εδώ πέρα την κυρία Ντανιέλα Γιούτο. Έχετε λοιπόν το λόγο για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Το θέμα αυτό θα Ήθελα να το ξαναθέσω, γιατί στο καλέ. Η κατάσταση ήταν ως εξή. Είχαν πάρα πολλά φορτηγά παρκαρισμένα και οι οδηγοί πέρασαν εβδομάδες, ε, μάλλον Σαββατοκύριακα ολόκληρα έτσι. Εσείς θα θέλετε έτσι, σε ένα τρέιλερ, σαν με ένα μικρό μπαλκόνι θα θέλατε να περάσετε σε αυτοκυριακό εκεί και αν όχι, γιατί δεν πληρώνετε καλύτερα τους οδηγούς σας για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά κομφόρ. Ε, ε, Η απάντησή μου είναι ότι στο Καλέτα τα Σαββατοκυριακά δεν είναι τόσο ωραία. Αλλά όσο υπάρχει ακόμα η ζούγκλα, ο κίνδυνο δεν είναι το σημείο συνάντηση ή το βενζινάδικο, αλλά το θέμα των μεταναστών, που προκαλεί πολλαπλά προβλήματα. Από την άλλη, αν η τρέχουσα νομοθεσία επιτάσσει χρόνο ανάπαυσης, τι να κάνουμε. Δεν έχουμε επιλογή παρά να περιμένουμε για να ξεκινήσει η επόμενη περίοδος οδήγησης και να μπορέσουμε να περάσουμε τη σειρά της μάχης σε ό,τι αφορά την σωστή αμοιβή. Μπορείτε να θέσετε το ερώτημα και σε μένα, αλλά όλοι στην Ουγγαρία θα ήθελαν να βγάζουν τόσα όσα στη Σουηδία. Αλλά υπάρχει απλά η υπηρεσία, ε, διαφορά της υπηρεσίας ε, στην Ευρώπη. Δεν φταίω γι' αυτό. Στην ε, εταιρεία μας οι οδηγοί βγάζουν τετραπλάσιο, πενταπλάσιο ποσό από τον ε, κατώτατο μισθό και αν τους ρωτήσετε με την αμοιβή τους είναι ικανοποιημένοι. Δεν ναι, έχετε άλλε ερωτήσει, κύριε Λουγκρίν. Έχετε και τρία δευτερόλεπτα ακόμα. Θα ήθελα να θέσω και μία ερώτηση προς ε, τα συνδικάτο από τη Δανία που αντιμετωπίζουν λίγο πολύ το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς στην Σουηδία. Ήταν χρήσιμη, μάλλον πιστεύετε ότι ήταν καλή για τις, ε, Ευρωπαϊκές, για τις Δανέζικες Υπηρεσίες Μεταφοράς ε, η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν σωστά κατάλαβα είναι η απάντηση. Το ερώτημα ήταν κατά πόσον ε, η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμαινε ότι έχουμε πιο πολλά ε, φορτηγά στην Δανία. Κοιτάξτε, κατά πόσο ήταν καλό για τον ε, δανέζικο κλάδο των μεταφορών, το διεθνή κλάδο. Ναι, μία φράση λέει ο Πρόεδρος για να απαντήσετε. Ναι, νομίζω ότι οι δανέζικες μεταφορές θεωρούν ότι υποφελήθηκαν. Για αυτούς ήταν καλύτερο. Αλλά ω συνδικάτο δεν μπορώ να πω ότι είμαστε κατά τη ενιαίας αγορά ούτε κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε απλά να υπάρχουν σωστοί κανόνε σωστέ συνθήκε εργασία. Και τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θέλουμε να είμαστε και σκλάβοι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρία λεπτά, η επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω ήδη λάβει αρκετέ απαντήσει στι προηγούμενε ανταλλαγέ, αλλά για τον κύριο Παρίγιο, εσείς θα ήσασταν υπέρ οι συνθήκες ε, οι εργασιακές ε, για τις χώρες υποδοχής να εφαρμόζονται από την πρώτη μέρα απόσπασης ε, και για να προστατεύσουμε πάντα τους εργαζόμενους που είναι και το πρώτο μας μέλημα μήπως θα ήταν θετικό να υπάρχει μια περίοδος μεταξύ δύο καμποτάς, μια περίοδος ξεκούρασης ναι Βεβαίω, εμεί στην ΕΤΕΦ θέλουμε η εφαρμογή να ισχύει από την πρώτη μέρα, άλλωστε αυτό ισχύει και σήμερα. Αυτό ισχύει σήμερα. Εφαρμόζεται από την πρώτη μέρα. Και βεβαίως η πρότασή μα είναι μετά από μια περίοδο καμποτάζ να υπάρχει περίοδος ξεκούραση. Προφανώς. Και να υπάρχει και ένα ενιαίο μέρο στην Ευρώπη γι' αυτό για να μην ε, γίνονται οι δηλώσεις ε, από εδώ και από εκεί να είναι ένα μέρος όπου θα μπορούν να βρουν οι επιθεωρητές οι Ευρωπαίοι στοιχεία και βεβαίως εδώ υπάρχει ένα αίτημα και των εργοδοτών που θέλουν όταν ελέγχουμε 100 οχήματα και που 70 ε, ε, είναι ε, νομότυπα να ελέγχονται τα υπόλοιπα 30 μόνο και να μην ε, σπαταλείτε χρήμα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί, έχουμε πάλι, γιατί έχει μπει η σημερινή το 2034 και όχι το 2022 από την Κομισιόν. Δεν φαίνεται να θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Η κυρία Λουκασένσκα έχει το λόγο. Δυόμιση λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και έχω κάποιες εξαιρετικές, ε, κάποιες ερωτήσεις να κάνω στην κυρία Μπερτούλα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το καμποτάζα, Όταν θα εξετάσουμε το καμποτάζ για την οδηγία, για την απόσπαση, κάθε οδηγός θα είναι ανεξάρτητος από το κράτος μέλος του. Και όλοι θα έχουν ε, την ίδια, τον ίδιο ρυθμό ορών. Γιατί υπάρχει τέτοια απροθυμία εναντί του καμποτάζ. Η Γαλλία πληρώνει τις ε, εταιρείε μεταφορικού μεταφορών από την Ανατολική Ευρώπη χαμηλότερες, ε, χαμηλότερους μισθούς. Γιατί δεν πληρώνουν με γαλλικούς όρους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο γι' αυτό. Και κάτι άλλο. Τα γαλλικά σούπερ μάρκετ, όπως για παράδειγμα το ΩΣΑ. Ε, κατακλείζουν την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι δική, δική ορία ανταγωνισμού αυτή. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Παρίγιο. Είσαστε κατά του να ξεκουράζονται και να κοιμούνται στο φορτηγό οι οδηγοί, γιατί δεν υπάρχει σωστή υποδομή στην παρούσα φάση. Και τα αγαθά τα οποία μεταφέρονται ενδεχομένω να είναι και επικίνδυνα. Θα φροντίσετε λοιπόν και θα ζητήσετε οι εταιρείε να εξοπλίσουν τις καμπίνες με κρεβάτια Πολλές οι ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να απαντήσω γρήγορα. Πρώτον, αν στη Γαλλία συνέβαινε ο οδηγός στα πλαίσια της απόσπασης να πληρώνεται λιγότερο από ότι ένας Γάλλος οδηγός, τότε αυτό θα αντιστοιχούσε σε απάτη. Αν λοιπόν συμβεί κάτι τέτοιο, μιλάμε για απάτη και δεν το δεχόμαστε προφανώ. Δεν μπορώ να συγκρίνω τα προϊόντα του οσών με του οδηγού, δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα, το για την ίδια κατάσταση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο λοιπόν γι' αυτό. Επίσης το ερώτημα είναι πολύ εύστοχο όμως το άλλο. Όταν μιλάμε για απόσπαση, τι κανόνες ακριβώς εφαρμόζουμε μετά την ε, διάσκεψη των Υπουργών της 23ης Οκτωβρίου είναι κάτι το οποίο θέλουμε να διευκρινίσουμε. Αν δούμε την οδηγία απόσπασης δεν έχουμε μόνο τους μισθούς, έχουμε και όλο το υπόλοιπο πλαίσιο πληρωμένες άδειες μεταποδοχών κτλ. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα δεν ισχύουν τα, ε, οι ίδιοι κανόνες για όλες τις χώρες. Όντως, ε, για τις διευκρινήσεις αυτές θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. Ο κύριος Παρίγιο, πολύ σύντομα, το ETF ε, δεν είναι κατά της ανάπαυσης στην καμπίνα της οδήγηση επειδή δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Είμαστε κατά της ανάπαυσης αυτής γιατί προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε σωστά τον κανονισμό. Έχει γίνει και μια προσφυγή μάλιστα και θα αποφανθεί πολύ γρήγορα ο Γενικό Αγγελέα του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κίνδυνο για τα εμπορεύματα, ναι, αλλά αυτό είναι ευθύνη τη επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή απαγορεύεται σε έναν οδηγό να εργάζεται κατά τη διάρκεια της ανάπαυσή του. Δεν μπορεί λοιπόν κατά τη διάρκεια τη ανάπαυση αυτή να προσέχει τα προϊόντα, γιατί θα φτάσει τότε σε εβδομάδα εργασία 90 ωρών, το οποίο είναι απαράδεκτο προφανώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει τώρα το λόγο για 2,5 λεπτά. Ναι, για την κυρία Μπερτελό. Ποιο είναι το per diem που, σας, που πληρώνουν του οδηγούς σας για το ξενοδοχείο και το ασφαλές πάρκινγκ. Στην συλλογική μας σύμβαση έχουμε την πληρωμή για την διατροφή και 56 ευρώ για τη διανυκτέρευση και για, τα, για τη διατροφή, ανάλογα με το αν είναι πρωινό ή μεσημεριανό, δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορώ να σας τα στείλω όμως τα στοιχεία αυτά. Εσείς ελέγχετε αν τους πληρώνουν, ε, δηλαδή τους παρουσιάζουν κάποια επόδειξη, κάποιο τιμολόγιο ή είναι απλό μέρος του μισθού. Ελέγχετε αν δαπάνησαν για αυτόν τον σκοπό. Ακούστε, είναι μια συλλογική σύμβαση που προβλέπει ότι είναι μια συνεισφορά του ε, εργοδότη στα ε, έξοδα μεταφοράς. Το ελέγχει η επιχείρηση, το ελέγχει και η επιθεώρηση εργασίας, διότι δεν υπόκειται ε, σε, ε, στις ε, εισφορές τις κοινωνικές. Οπότε ελέγχεται ιδιαίτερα. Δεύτερο ερώτημα. Είδα εγώ στην παρουσίασή σας ότι έχετε χωρίσει τους οδηγούς και, τα, και τις ποσότητες ε, μεταξύ εθνικών και αλλοδαπών έχετε κάπου μια κατηγορία για τους Ευρωπαίους ε, ε οδηγούς και τους μη Ευρωπαίους ε, ή τους βάζετε όλους μαζί. Όχι, δεν έχουμε κάνει διαχωρισμό αυτόν αναοδηγό, αλλά ανασημαία ε, και στην πρώτη είναι όλοι μαζί στην πρώτη διαφάνεια. Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι Μαροκινοί, μπορεί να είναι Ουκρανοί, Ισπανοί, όλοι το ίδιο. Όχι, όχι. Εδώ μιλάμε για ευρωπαϊκή σημαία. Έχουμε πολύ πιο λεπτομέρειε διαφάνειε του ή άλλου πάντω για την κάθε χώρα ξεχωριστά και μπορούμε να σα τι προμηθεύσουμε. Το, η Εθνική Οδική Επιτροπή είναι που τα καθορίζει αυτά. Ε, είπατε για την επιστροφή στο σπίτι ότι λέτε ότι αυτό μπορεί να είναι παγίδα διότι δεν υπάρχουν μέτρα που να το, ε, καθιστούν ελέγξιμο. Ε, γιατί είδου μέτρα μιλάτε, γιατί μέτρα μιλάτε δεν με ρωτήσε κανείς τίποτα για την επιστροφή. Ο κύριος Παρίγιο, στον κύριο Παρίγιο απευθύνομαι για την επιστροφή. Ναι, ακούστε, σήμερα στην πρόταση που έχει υποβληθεί αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά ποιο είναι ο που δίνεται στην έδρα, στον, στον, τόπο διαμονής, εν περιπτώσει, συγγνώμη, Οπότε είναι κάτι που μπορεί να γίνει και να μην γίνει. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να υποχρεώσουμε κάποιον να επιστρέψει ε, ενώ θα τον πιέζουμε μετά από τέσσερις εβδομάδες για να πει, ξέρεις, ε, να ξέρετε, να το πούμε, ξέρεις ξαφανίσου για μια εβδομάδα και επέστρεψε μετά για να λάβεις ε, καθήκοντα. Όχι, δεν ρωτάω για την πρόταση, ρωτάω για τη δική σας θέση, έτσι ώστε η επιστροφή να είναι δικαίωμα των εργαζομένων. Ξέρετε ότι ο όσου είναι περιφερειακού εργαζόμενο, αυτό είναι ένα πραγματικό αίτημα. Η δική σα θέση λοιπόν ε, για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε το κείμενο στη επιστροφή να είναι ένα δικαίωμα το οποίο να ελέγχεται. Όχι τι νομίζετε για τη θέση τη Κομισιόν. Ε, ναι, μια φράση κύριε Παρίγιο. Να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ελέγχου σοβαρό. Σήμερα δεν υπάρχει απολύτω τίποτα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Η κυρία Φώστερ έχει το λόγο. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και συγγνώμη, κάποιε από τι απόψει δεν τι άκουσα νωρίτερα, δεν ήμουν εδώ. Συγγνώμη να επαναλάβω ερωτήσει. Τα μέλη του πάνελ συμφωνούν σε σχέση με την έκθεση της Κομισιόν για την συμπερίληψη των οχημάτων κάτω 3,5 τόνων εγώ δεν είμαι υπέρ του να διαβρεθεί το πεδίο εφαρμογή και να καλύψει και αυτά τα οχήματα. Δεν τώρα μιλάω όταν μιλάμε για μικρέ ε, ε, αποστάσει. Επίση υπάρχει ένα θέμα οικονομικό για αυτά τα μικρά οχήματα. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι έχουν να πούν τα μέλη του πάνελ. Αν συμφωνούν με τη δική μου θέση ε, και αν θεωρούν ότι πρέπει ε, ε, να μην αλλάξει το πεδίο εφαρμογής. Ναι, για να απαντήσω στο ερώτημα, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Θέλουμε να συμπεριληφθούν τα οχήματα κατά από 3,5 τόνου, να συμπεριληφθούν με προποθέσει πρόσβαση βέβαια, ε, που να είναι λίγο πιο χαλαρέ σε σχέση με αυτά που ισχύουν για τα μεγαλύτερα οχήματα. Εμεί είμαστε σαφώ υπέρ τη συμπερίληψη των οχημάτων κάτω των 3,5 τόνων. Συμφωνούμε απολύτω. Και για την πρόσβαση στην αγορά. Ε, δεν χρειάζεται πια να μιλάμε για τον ΝΑΖ από τη στιγμή που κάνουμε διεθνείς μεταφορές, όποιο και αν είναι το τονάζ, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην, ε, στο επάγγελμα και να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες. Να συζητήσουμε το πώς μπορεί να γίνει αυτό, βέβαια, ανάλογα με το, το, το τα οχήματα, αν είναι 40 τόνων ή κάτω από 3,5 τόνων, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι όλοι να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Εγώ μίλησα για λιγότερο από 3,5 τόνους. Όχι 31, Α, μπορεί να ήταν η μετάφραση. Α, μάλιστα, ευχαριστώ. Δύο ακόμα σύντομα σημεία. Ο ορισμός της, διεθ, της διεθνούς ε, μεταφοράς ε, για τις αυτό καλύπτει τις μεγάλες ε, εκδηλώσεις, τις αθλητικές, υπάρχουν περιορισμοί από αυτού και αυτό μπορούμε να, να το αποφύγουμε εάν τους ορίσουμε για τις διεθνείς μεταφορές. Πώς σας φαίνεται αυτό. Λοιπόν, με την ευκαιρία πρέπει να προσέξουμε να χρησιμοποιούμε ορισμού. Εγώ ακούω κάποια πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ καθόλου. Ε, όταν έχουμε μια μεταφορά από την χώρα Α προ τη χώρα Β την οποία εκτελεί μια χώρα Γ, αυτό δεν είναι διεθνέ ε, ε, διεθνής μεταφορά που ο κάνει ό,τι θέλει. Όχι, εφαρμόζεται, ε, εφαρμόζεται ο μισθό της χώρας Α ή τη χώρα Β και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι Τέλειωσε ο χρόνο. λυπάμαι, συνεχίζουμε. Ο κύριος Βαν Μίλτεμπεργκ έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, προ τον κύριο Σχίπερ, λέτε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την τήρηση των κανόνων τι σκέφτεστε για να κάνετε καλύτερη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πέρα από τον τα e ταφογράφο. Πιστεύετε ότι έχουμε κάποια δυνατότητα να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κάποιες τροπολογίες και πείτε μας τι σκέφτεστε. Η απάντηση Ε, ακούσαμε κάτι για την πρόσβαση στα εθνικά μητρώα των ε, υπεύθυνων ε, επιτήρησης. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι τα τρέχοντα στοιχεία τήρησης. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει μετά από επιβολή κύρωσης και πρόστιμο και αυτό μπορεί να πάρει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ θέλω τα σύγχρονα. Τα, τα πιο τελευταία στοιχεία για τις εταιρείε που δεν τηρούν ε, τους κανόνες. Αυτό θα χρειαζόμουν. Μάλιστα. Και συμφωνείτε ότι θα πρέπει να βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις σε ό,τι αφορά το μορφότυπο, για παράδειγμα, των δεδομένων, προκειμένου να είναι επίκαιρα. Ναι, απολύτως. Είναι καλή ευκαιρία αυτή, λοιπόν, για μας τους νομοθετές να καταθέσουμε νομοτροπολογίες. Ε, Προς τον κύριο Παρίγιο, μια ερώτηση. Δεν έχω καταλάβει καλά. Συμφωνείτε για την εισαγωγή, την ταχεία ε, εισαγωγή των ε, έξυπνων εφιών ταχογράφων. Απάντηση. Ναι, το συντομότερο δυνατόν. Τον Ιούνιο του 2019, μα γίνεται. Και την ίδια ερώτηση για τον κύριο Α, από την Ουγγαρία. Θέλετε να είναι ταχεία η εφαρμογή των έξυπνων ε, ε ταχογράφων. Εμείς ε, διαφωνούμε με την νομοθεσία, όχι με το τεχνολογικό σκέλος. Μάλιστα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για μας ε, ως νομοθέτες. Ευχαριστώ πέρα. Ευχαριστούμε κύριε Φαν Μίτλμπεργκ. Ο κύριος Κόχ. Πώς ε, ε, εκτιμάτε την, ε, επιπτώσεις του παράνομου καμποτάζ και τι μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μια ρεαλιστική λύση ο κύριος Σκύπερ. Δεν έχω καμία ιδέα για το ποσοστό, να σας πω την αλήθεια. Αυτό εξαρτάται και από το πώς ε, προσμετρούμε. Και δεν έχουμε και μέσα να κάνουμε τον έλεγχο. Θα πρέπει φυσικά να θέσουμε και προτεραιότητες, το για παράδειγμα τις χώρες Μπενελούξ, μεταξύ των χωρών Μπενελούξ το καμποτάζ είναι ελεύθερο. Δεν έχουμε λοιπόν ιδιαίτερη εμπειρία. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για το ποσοστό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να το εκτιμήσω. Σας ευχαριστώ κύριε Παριά. Αν θέλετε να... Αν θέλετε να κρατήσετε ένα κατάλογο προτεραιοτήτων για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους ε, συνθήκες εργασίας, ποια τρία μέτρα θα ήταν στην κορυφή των προτεραιοτήτων σα. Πρώτο μέτρο, η εφαρμογή, η άμεση εφαρμογή των εφιών ε, ταχυγράφων. Το Εθνικό Μητρό, το οποίο, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες οι υπηρεσίες ελέγχου, προκαταρτική δήλωση για τις μεταφορές και μια ευρωπαϊκή υπηρεσία η οποία θα ελέγχει επίσημα και όχι σε εθελοντικό επίπεδο όπως το ECR. Άρα να χορηγήσουμε τα εργαλεία τα οποία χρειάζεται κάθε εταιρεία προκειμένου να έχει ίσους όρους ανταγωνισμού και το ίδιο και για τους εργαζόμενους επίσης να έχουν ίσους όρους εργασίας ίση αμοιβή για την ίδια δουλειά σε κάθε χώρα. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία είναι τα πιο σημαντικά και τα πιο γρήγορα και τα πιο καταπήγοντα αν θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Άντερσον, παρακαλώ στον Πορτογάλο εμπειρογνώμονα για τα οχήματα σε ό,τι αφορά τα, την ενοικίαση φορτηγών. Τι χρησιμοποιείται και αν ναι, γιατί και αν όχι επίσης γιατί. Κατά δεύτερον πιστεύετε ότι το μέτρο αυτό που προβλέπεται στην οδηγία του 2016 που επιτρέπει την ακόμα μεγαλύτερη απελευθέρωση από κάποια κράτη-μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε και τότε. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπήρχαν κοινά πρότυπα παρά να επιτρέπουμε κάποιους διαφορετικούς βαθμούς απελευθέρωσης στις αγορές. όλες οι υπηρεσίες στην Πορτογαλία, οι μεγάλες ε, ε, εταιρείε τουλάχιστον, έχουν όντως ε, ενοικιαζόμενα φορτηγά και μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ίδιο κεφάλαιο ή να δανειστεί για να χρηματοδοτήσει αυτές τις ενοικιάσεις. Και αυτό επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίε και κάποια από αυτά τα φορτηγά χρησιμοποιούνται και για κατοκαμποτάζ. Τώρα, η απελευθέρωση του κλάδου συμπεριλαμβανομένης και της απελευθέρωσης των ε, ενοικιαζόμενων οχημάτων για εταιρείε οι οποίες ε, μεταφέρουν δικά τους προϊόντα. Θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι οι λιγότερο αποδοτικοί μεταφορείς που κάνουν ε, ένα ταξίδι άδειοι, μπορούσαν να συνεχίσουν. Εμείς θέλουμε να επικρατήσουν όμως οι πιο αποτελεσματικοί, οι πιο αποδικοί μεταφορές για να, μετα... να περιορίσουμε και το αποτύπωμα του ανθρακά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε τέτοια ενοικιαζόμενα φορτηγά, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Και θα πρέπει να πετύξουμε προσοχή. Δεν θέλουμε υπερβολική απελευθέρωση σε ό,τι αφορά το leasing των φορτηγών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κλούντορ, έχει το λόγο. Δύο μισή λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απευθύνομαι καταρχάς στον καθηγητή κύριο Πορκόφσκι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη μελέτη σας. Πολλά αριθμητικά δεδομένα θα πρέπει να τα μελετήσουμε λίγο πιο προσεκτικά. Μια διευκρίνηση θα ήθελα αναφερθήκατε σε περιφερειακές και κεντρικές χώρες. Και είπατε ότι οι περιφερειακές χώρες έχουν ε, μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες θα επηρεαστούν τελικό περισσότερο από τις κεντρικές χώρες που έχουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις με περισσότερα κεφάλαια. Άλλοι αναφέρθηκαν στη συνέχεια σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και ωστόσο τόσο πολύ σε περιφερειακές χώρες. Στη μελέτη σας επικεντρωθήκατε κυρίως στην Πολωνία. Πώς μπορούμε να προβάλλουμε τα δεδομένα αυτά και στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε. Κοιτάξτε, δύο μελέτες γίνανε. Η πρώτη είχε να κάνει όντως με την Πολωνία όπου σας έδωσα συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα για τις επιπτώσεις, ενώ η δεύτερη ήταν μια οικονομικομετρική μελέτη, η οποία ήταν πανευρωπαϊκή και αναφερόταν όντω σε κεντρικές και περιφερειακές χώρες. Τα συμπεράσματα είχαν να κάνουν με αυτή την οικονομικομετρική μελέτη. Όσον αφορά τις περιφερειακές χώρες, δεν αναφέρομαι μόνο στις 13 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις 15. Εκεί βάζω λοιπόν και την Πορτογαλία και την Ιρλανδία λοιπόν, η οποία θα είναι ακόμα πιο απόκεντροι. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ακόμα ερώτημα προς τον κύριο Βιλάτσεν. Α, χρησιμοποίησατε τον όρο «καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης» μιλώντας για το χρόνο ανάπαυσης στον θάλαμο οδήγησης. Πώς μπορούμε αυτό από νομοθετικής πλευράς να το συμπεριλάβουμε, γιατί καταλαβαίνετε από τον ένα μιλητή στον άλλον, από μια χώρα στην άλλη, μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εννοούσα είναι ότι στα πλαίσια της αγοράς εργασίας θα πρέπει να μπορεί κανείς να εξορροπεί προσωπική και επαγγελματική ζωή. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου το ότι ε, ένας οδηγός ο οποίος καλείται να ζήσει σε δύο τετραγωνικά μέτρα σε, για 20 μέρες το μήνα, πρέπει να μπορεί ο άνθρωπος αυτός να αναπέβεται λίγο περισσότερο και με συνθήκες πιο αξιοπρεπείς. Όχι δηλαδή αναγκαστικά μόνο μέσα στο φορτηγό, θα πρέπει στα πλαίσια της προβλεπόμενης για ανάπαυσης να μπορεί να επιστρέφει και στο σπίτι του. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε. Κύριε Έρτουκ, έχετε εσεί το λόγο για δυόμιση λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ξαναθέσω μια ερώτηση προ τον κύριο Λάικο. Κύριε Λάικο, άκουσα αυτά που είπατε ω τώρα. Αυτό που βγάζω συμπέρασμα είναι ότι η Ουγγροί οδηγεί με ουγγρικούς μισθούς και ουγγρικά φορτηγά κάθε τέσσερις εβδομάδες ε, πρέπει να πάνε στην Ουγγαρία, στην πατρίδα τους και παράλληλα Είπατε και σε απάντηση στον κύριο Φαντενκάμπ, αν δεν κάνω λάθος, ότι η δουλειά, ότι οι οδηγοί τουλάχιστον ε, για τη δουλειά τους ε, βρίσκονται συχνά στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Γιατί λοιπόν απασχολείτε τους ε, εργαζόμενούς σας, τους οδηγούς σας, σύμφωνα με τους γαλλικούς, τους γερμανικούς όρους. Ίσως να υπάρχει κάποια παρανόηση στα πρέπει να το αφαιρέσουμε αυτό από τον, τον χρόνο ξεκούραση. Κάθε 9 μέρες υπάρχει ένα χρόνο ξεκούραση. Κάθε 9 ώρες υπάρχει ξεκούραση. Το καλέ λοιπόν, όχι, όχι, δεν μιλάω για τον χρόνο εργασία, Εγώ λέω, προσπάθησα να εξηγήσω ότι αυτό, αυτό που είπατε εσεί νωρίτερα. Είπατε, ο Ούγγρος οδηγός ε, έχει τη δουλειά του στη Γερμανία, στη Γαλλία και λέτε ότι αυτό δεν είναι καμποτάζ. Ακολουθώ λοιπόν τη λογική σας. Αυτό σημαίνει ότι ο Ούγγρος οδηγός με ουγγρικούς κανόνες, με ουγγρικά πρότυπα, οδηγεί στην Ευρώπη και επιστρέφει μετά από τρεις εβδομάδες στη χώρα του στην Ουγγαρία. Έτσι. Αν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα, γιατί χρησιμοποιείτε, ε, χρησιμοποιείτε τα γερμανικά και τα γαλλικά πρότυπα. Εγώ προηγουμένω είπα τέσσερι εβδομάδε είναι το maximum και το μέσο, μέσο όρο στο εξωτερικό και τον Ούγγρο οδηγό στις εταιρείε μας είναι 2,5 εβδομάδες. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Σε αυτό το ταξίδι ο οδηγός ε, δεν αφορά μόνο αυτή η μεταφορά ουγγρική, ουγγρική μεταφορά, αφορά ευρωπαϊκή. Δεν είναι όμως περίπτωση καμποτάζ. Ναι, συγγνώμη που διακόπτω, δεν θα έχω και χρόνο. Για άλλη μια φορά. Οι προδιαγραφές που ακολουθούνται, τα πρότυπα, είναι τα ουγγρικά. Είπατε όμως ότι εργάζονται κυρίως εκτός Ουγγαρίας. Είναι Ουγγρι, Ούγγροι οδηγοί, Ούγγρικα φορτηγά που όμως δραστηριοποιούνται εκτός Ουγγαρίας. Επιστρέφουν από τρεις εβδομάδες. Εφόσον είναι έτσι τα πράγματα και αυτό είναι το επιχείρημά σας, πώς εξηγείτε και γιατί δεν χρησιμοποιείτε τις προδιαγραφές ε, του τόπου όπου εργάζονται στη Γαλλία, στη Γερμανία. Ναι, το θέμα είναι ποιε θα είναι οι προδιαγραφέ, διότι σε τρει εβδομάδες ο μέσος οδηγός ε, θα περάσει από όλε τι χώρε της Ευρώπης. Ε, δηλαδή κάθε δύο μέρες αλλάζει χώρα. Προσπαθείτε να καταλάβετε τι θα γίνει. Θα έχει ένα διαφορετικό συμβόλαιο για την κάθε χώρα από την οποία περνάει. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ναι, αλλά το πάλι στο γραφειοκρατικό τώρα. Δεν απαντήσατε όμως το βασικό. Λοιπόν, μια τελευταία προσπάθεια σε μια φράση. Περιμένω τη μετάφραση. Μα δεν υπάρχει ερώτηση όμως να υπάρξει μετάφραση. Ποιο είναι το ερώτημα. Νόμιζα ότι είχα απαντήσει στο ερώτημα. Ε, εντάξει. Ξαναρωτήστε πάντως αν θέλετε. Η κυρία Ροβονταλόν για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Το ερώτημά μου αφορά τον κύριο Μπορκόφσκι. Ο κύριος Μπορκόφσκι μας, έκανε μια παρουσίαση των μελετών του στην Πολωνία. Θέλω να ζητήσω, να ρωτήσω κάτι για τους ε, οδηγούς στην Πολωνία και ιδιαίτερα στα διοδρομία τους. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η διάρκεια της σταδιοδρομίας ενός ε, οδηγού έτσι όπως το περιγράψατε, με μικρή, μικρό χρόνο ξεκούρασης. Ε, πόσοι, πόσες ε, διακοπές έχουν, πόση άδεια έχουν, πληρωμένη άδεια ετησίως, τι συμβαίνει όταν ε, είναι ασθενής, τα αναλαμβάνει τα έξοδα ε, η εταιρεία τους και για ποιο ύψος έχουν δικαίωμα στη σύνταξη και ποιο είναι επίσης το ποσοστό ατυχημάτων με βάση τη μεγάλη διάρκεια εργασίας ε, αυτών των οδηγών. Έχετε απαντήσει τα ερωτήματα αυτά. Ακούστε για τον Πολωνό οδηγό, τον Πολωνό εργαζόμενο ε, εφαρμόζεται η πολωνική νομοθεσία. Όλα όσα ρωτήσετε αφορούν την πολωνική νομοθεσία. Σύνταξη, ε, ε, τα, η άδεια, τα όποια ωφελήματα, τη υγειονομική κάλυψη. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Εφαρμόζεται αυτό που εφαρμόζεται για όλους τους λοιπούς εργαζόμενους στην Πολωνία. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ε, ποια είναι τα στοιχεία αυτά. Δεν είμαι εργατολόγος, δεν ξέρω τα ακριβή στοιχεία, αλλά δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο στην Πολωνία. Τώρα για το ποσοστό ε, ατυχημάτων, συγγνώμη, συγγνώμη, εάν μου λέτε ότι τα δικαιώματα του ε, οδηγού είναι τα ίδια με αυτά οποιοδήποτε εργαζόμενου, δηλαδή ο χρόνος εργασίας που του οδηγού είναι ο ίδιος με το χρόνο εργασίας του εργαζόμενου, του οποιοδήποτε εργαζόμενου, υπάρχει ξεκούραση το Σαββατοκύριακο ή εργάζεται τρεις εβδομάδες. Ακούστε, για μιλάω για τους οδηγούς στην Πολωνία. Οι οδηγοί στην Πολωνία και οι οδηγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν τους κανόνες που προβλέπει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είπατε για τη σύνταξη και άλλα πράγματα εσείς. Αυτά τα ρυθμίζει η πολωνική νομοθεσία. Τώρα δεν μπορώ να το πω τα στοιχεία διότι δεν είμαι εργατολόγο. Επαναλαμβάνω. Δυστυχώ δεν μπορώ να σας συνδράμω εδώ. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Τρία λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ναι, καλημέρα σας κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος, διότι εδώ βρισκόμαστε να ακούσουμε τον κλάδο. Θα είμαι σύντομος πέντε σημεία. Πρώτον, μπορείτε να μιλήσετε γαλλικά εφόσον το επιθυμείτε. Έπρεπε να υπήρξε μεγαλύτερη διαβούλευση πριν υποβληθεί η πρόταση η νομική. Κάποια στιγμή όμως έπρεπε να γίνει και η πρόταση. Εμείς αναλάβαμε την ευθύνη μας. 31 Μαΐου υποβάλαμε την νομική πρόταση για να ξεκινήσει και η συζήτηση στο Συμβούλιο και, με το, στο Κοινοβούλιο. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει ένα πακέτο όπου υπήρξε διαβούλευση, ε, είναι αυτό. Δημόσια διαβούλευση, ε, διασκέψεις ε, και βεβαίως πάρα πολλές συναντήσεις ε, με τους εμπλεκόμενους φορείς. Δεύτερο θέμα και ελπίζω έτσι να ικανοποιηθεί ο κ. Βαντενκάμπ για την ψηφιοποίηση. Ακούστε, η ψηφιοποίηση είναι πολύ σημαντική βεβαίως, όχι μόνο για να βελτιωθούν οι έλεγχοι, αλλά και για να μειωθεί η επιβάρυνση από τον έλεγχο σε όλους. Έχουμε κάνει προτάσεις, έχουμε ετοιμάσει τον κανονισμό για τον ταχογράφο, θα επιβάλλουμε ε, το ECMR Βεβαίω, αν μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η πρόταση τη Κομισιόν, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγο πάντω τα κράτη-μέλη ή το Συμβούλιο να μην ακολουθήσουν αυτήν την οδό. Τρίτο σημείο, το κόστο τη νομοθετική πρόταση ε, για τον τομέα, για τον κλάδο. Βεβαίω πολύ σημαντικό το θέμα. Η πρόταση πρέπει να είναι ισορροπημένη, πρέπει να είναι αναλογική εγώ θα έλεγα ότι η εσωτερική, αγορά ε, σίγουρα υπάρχει μεγάλο κόστο για τον κλάδο, αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί το σημείο ισορροπία του στόχου τη εσωτερική αγορά, να μειωθεί το κόστο για τον κλάδο με τον άλλο στόχο, που είναι να βελτιωθεί οι, κοινωνική, οι κοινωνικές συνθήκες για τους εργαζόμενους και τους οδηγούς. Και ένα στοιχείο σε ό,τι αφορά το κόστος για τον κλάδο τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την απόσπαση των εργαζομένων και τη σχετική οδηγία που συζητήθηκε επί μακρόν. Σήμερα, στη λέξη Specialis, εμείς προτείνουμε συγκεκριμένους κανόνες ακριβώς για να προσαρμόσουμε τα μέτρα ελέγχου στις ε, οδικές μεταφορές διότι έχει μια ιδιαίτερη φύση αυτός ο κλάδος. Τέταρτο σημείο, η υπηρεσία, ο οργανισμός η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα στην πρόσθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση μια τέτοιας υπηρεσίας. Βεβαίως γνωρίζετε ότι ο πρόεδρος Γιούγκερ έκανε μια ανακοίνωση στην ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθέστησε σαφές ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία εργασίας ξέρω ότι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης ε, ασχολούνται με αυτό και τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών θα συνεχίσει να συμμετέχει ε, ενεργά στην προπαρασκευή αυτής της πρότασης. Δηλαδή εμείς στην DG Move ε, θεωρούμε ότι αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Και θα κλείσω για να απαντήσω και στον κύριο Λούγκρεν που λέει κατά πόσο θα πρέπει ενδεχομένως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει καταστρέψει τον τομέα των μεταφορών. Ε, ακούστε, εγώ θα σας πω βέβαια ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως φαντάζεστε. Αντιθέτως, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχε, θα συνεχίζαμε να ρυθμίζουμε τις μεταφορές με ένα σύστημα ποσοστώσεων. Θα υπήρχε θα υπήρχε θα υπήρχαν σύνορα, ουρές στα σύνορα, εμείς λοιπόν στην Κομισιόν θεωρούμε ότι η εσωτερική αγορά έχει στεφθεί από επιτυχία, πρέπει αυτή την επιτυχία να την διαφυλάξουμε, αλλά επίσης αυτή η εσωτερική αγορά πάει χέρι-χέρι με μια ισχυρή κοινωνική πολιτική, μια ισχυρή κοινωνική διάσταση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τη συζήτηση αυτή την υποδομητική Σήμερα ήταν μια σημαντική συνεισφορά στις εργασίες μας για το πακέτο για την κινητικότητα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορέσαμε να, ακούσαμε, να ακούσουμε τις απόψεις για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Παρακαλώ, παρακαλώ ένα χειροκρότημα για όλους τους παρεμβαίνοντες που ήταν εδώ εδώ και δύο ώρες και απαντάνε σε ερωτήσεις σας. Και συνεχίζουμε αύριο στις 9.30 δεύτερο πάνελ για την ε, τιμολόγηση την οδική. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κάνουμε ένα διάλειμμα για 7 λεπτά και στη συνέχεια έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε 7 λεπτά.